Thank you very much for coming so early. Κυρίες και κύριοι, ε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε τόσο νωρίς ε, παρά την ε, κοσμική ζωή που μπορεί κανείς να απολαύσει στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και ξεκινάμε με το σημείο που βλέπετε στην ημερησία διάταξη. Κάθε χρόνο παρουσιάζουμε μια γενική επισκόπηση που αφορά στην ε, πολιτική ασφαλείας και εξωτερική πολιτική. Και ήθιστε πρόεδρος αυτής της έκθεσης να είναι ο το πρόεδρος ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε προετοιμάσει αυτήν την ε, έκθεση. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα επεξεργαστήκαμε ένα πρώτο έγγραφο εργασίας το οποίο έχει κατατεθεί προς συζήτηση γιατί δεν έχει λάβει ακόμα την τελική του μορφή. Υπάρχει προσπάθεια να δούμε τα σημαντικότερα θέματα και να εξετάσουμε την κατάσταση σε διάφορες χώρες του κόσμου. Θα χαιρόμουν λοιπόν πάρα πολύ αν ε, οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, κυρίως αυτοί ε, μπορούσαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, ε, μπορούσαν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους και αν θέλουν και κατά τις επόμενες μέρες και εβδομάδες για να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή, την επισκόπηση. Σας καλώ λοιπόν θερμά, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, να μου αποστείλετε το συντομότερο δυνατόν τις ε, παρατηρήσεις έτσι ώστε όταν θα συντάξω την τελική έκθεση να μπορώ να λάβω υπόψη μου και τις δικές σας απόψεις. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε νέες εξελίξεις τόσο όσον αφορά τα εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τις εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό αφενός και αφετέρου για να δούμε τα βασικότερα θέματα που οφείλει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να βελτιώσει τις δικές δομές. Τα τελευταία 4-5 χρόνια ασχοληθήκαμε με την ε, σύσταση της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Εκεί τα καταφέραμε αρκετά καλά, αλλά βέβαια θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι προφανώς και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης εξακολουθεί να έχει ακόμα αδυναμίες που πρέπει να καλυφθούν τόσο όσον αφορά την ίδια την υπηρεσία όσο και όσον αφορά την δυνατότητα πολιτικής τοποθέτησης ε, των αντιπροσωπιών στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα. Επίσης πιστεύω ότι οφείλουμε να ε, διαπιστώσουμε ότι ως προς τις ε, συνέργειες τις οποίες ε, συζητήσαμε χθε με την κυρία Μογκερίνη, στον τομέα αυτό οφείλουμε να δραστηριοποιηθούμε. Αν έχετε την καλοσύνη, εσείς εκεί, σας παρακαλώ κύριε, να ολοκληρώσετε τη συζήτησή σας. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι οι συνέργειες που αφορούν στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης και που επίσης αφορούν και στη θέση της ε, ΥΠΑΤΣ εκπροσώπου που είναι και αντιπρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωπος του Συμβουλίου, αυτές οι συνέργειες αυτή τη στιγμή δεν έχουν επιτευχθεί. Βεβαίως ε, εν μέρη διότι η υπηρεσία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά σε κάποιο βαθμό αυτό οφείλεται και στο ότι ε, δεν υπάρχει ακόμα η απαραίτητη πολιτική βούληση. Η ύπατη εκπρόσωπος ακόμα δεν έχει μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντά της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατ' ουσίαν δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε μία συνεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό οφείλεται και στη διένεξη με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία ακόμα δεν έχει ούτε καν επίτροπο, κάτι το οποίο διαπιστώνουμε ε, να έχει συνέπειες ε, σε, πολλές, ε, σε πολλούς Βλέπουμε ότι η Μεγάλη Βρετανία ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της και ίσως αυτό να οφείλεται βέβαια σε μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση. Βλέποντας το πρόσωπο του Τζόφρι βλέπω ότι χαίρεται για όλα αυτά, δεν τον βλέπω στενοχωρημένο. Όμως εφόσον υπάρχει αυτή η βρυβιακή κατάσταση ότι ε, πολλά θέματα της εξωτερικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής, ε, δηλαδή η πολιτική γειτονία, η πολιτική διεύρυνση, η εμπορική πολιτική, ε, όλες αυτές οι πολιτικές εμπίπτουν σε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δηλαδή καταλήγουμε στο ότι αυτό το αποτελεσματικό εργαλείο δεν χρησιμοποιείται, άλλα θέματα αποδίδονται σε διακυβερνητική συνεργασία. Αν θέλουμε όμως να έχουμε μία ολοκληρωμένη τοποθέτηση πρέπει όλα αυτά να τα συγκεράσουμε. Γι' αυτό λοιπόν υπήρξε, καταλήξανε στο ότι θα υπάρχει ένα άτομο το οποίο θα τα αναλαμβάνει όλα αυτά υπόψη του είναι εκείνο το οποίο θα τοποθετεί το πλαίσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνει τη σύζευξη ανάμεσα στη διακυβερνητική συνεργασία και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό όμως πρέπει να το επιτύχουμε αν θέλουμε να έχουμε και μια αποτελεσματική πολιτική. Και ε, θέλω όλα αυτά να σας τα εξηγήσω όλες. Βλέποντας ότι αυταρχικά καθεστώτα όπως παραδείγματος χάρη αυτά της Ρωσίας ή της Κίνας εφαρμόζουν αν θέλετε μία συμπαγή πολιτική, δηλαδή ακόμα και οι πιο μικρές αποφάσεις των χωρών αυτών που λαμβάνονται σε επιχειρησιακό επίπεδο, με μονομένες επιχειρήσεις δηλαδή από αυτές τις χώρες, οι αποφάσεις που λαμβάνονται εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική. Άρα δηλαδή εμείς στην περίπτωση αυτή είμαστε σε μειονεκτική θέση. Γιατί εμείς είμαστε σε μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία που έχουμε ελεύθερες επιχειρήσεις που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους περί και άλλες με καθαρά ελεύθερα και δημοκρατικά κριτήρια. Αλλά για δέστε που φτάνουμε στον τομέα της ενέργειας. Ίσως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια ενιαία εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι εφικτό. Αυτό σημαίνει ότι και στον πολιτικό τομέα πρέπει να υπάρξει σύζευξη των διαφόρων απόψεων για να μην υπάρχουν αντιφάσεις. Και επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτές ε, οι αντιφάσεις, το σημαντικότερο είναι, όπως σας είπα, να γνωρίζουμε ότι επειδή οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, ε, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης καλείται όλα αυτά να τα συγκεράσει, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως. Ε, η ε, ύπατη εκπρόσωπος της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης νομίζω ότι τα έχει όλα αυτά υπόψη αλλά πρέπει και εμείς να τη βοηθήσουμε για να επιτύχει το στόχο της. Και για να γίνει αυτό προτείνουμε μία σειρά οργανωτικών μέτρων γιατί πραγματικά υπάρχει μια αδυναμία, μια δυναμία που δεν έχουμε μπορέσει να την ε, εξαλείψουμε ούτε καν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την κρίση του Σαντέρ το 1999 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, κατέληξαν σε έναν τέτοιο ε, κανονισμό που είναι τόσο περίπλοκος ε, και ιδιαίτερα χρονοβόρος. Ε, αυτό ισχύει και για την εσωτερική πολιτική. Όμως αυτός ο χρηματοδοτικός κανονισμός ο οποίος είναι εκείνο που ισχύει και για βοήθεια στο εξωτερικό, αν αυτή η βοήθεια δεν χορηγείται έγκαιρα, προφανώς και πρόκειται για διασπάθηση χρήματος. Σήμερα μιλάμε για διάφορα πράγματα και ουσιαστικά τα χρήματα τα διαθέτουμε μετά από ένα-δύο χρόνια. Ε, τότε τι νόημα έχει αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά παραδείγματα για το πώς ε, μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο, αλλά εκείνο που είναι απαραίτητο να είμαστε αποτελεσματικοί και ως εκ τούτου καλούμεθα να λάβουμε μία σειρά μέτρων. Νομίζω λοιπόν ότι από αυτού είναι απαραίτητο να υπάρχει μία σε συζήτηση και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών για να αλλάξει η κατάσταση και επίσης για να μπορέσουμε να διευρύνουμε το πεδίο δράσης της ΥΠΑ της εκπροσώπου ε, σε θέματα εξωτερικής ε, πολιτικής. Άρα δηλαδή αυτά ισχύουν για την, για την πολιτική γενιτονίας και για πολλές άλλες ε, πολιτικές. Το δεύτερο θέμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι το εξής ότι όσον αφορά τα κράτη-μέλη χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους και πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν με τη σχετική συνθήκη να στηρίζουν ενεργά και να δείχνουν πίστη και αφοσίωση στην εξωτερική πολιτική. Και από αυτού πρέπει να σας πω ότι έχω πολλές αμφιβολίες. Εγώ φοβάμαι ότι κάθε υπουργό εξωτερικών κάνει μόνος του τα ταξίδια του, προβαίνει σε κάποιες ε, συμφωνίες και αν τα δει κανείς ε, απ' έξω όλα αυτά είναι σε αντίφαση με τα συμπεφωνημένα. Για μένα εκείνο που έχει σημασία είναι λόγω των τελευταίων και πρόσφατων εξελίξεων οφείλουμε να επιληφθούμε συγκεκριμένων πραγμάτων. Εδώ λοιπόν πρόκειται για το εξής, να αναπτύξουμε δράσεις που θα βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Αυτό να διασφαλίσουμε στην Ευρώπη και να προσπαθήσουμε να το επιβάλλουμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχει κατάσταση. Ε, διεξάγεται μια συζήτηση που δεν αφορά μόνο στην Ουκρανία. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι με την συμφωνία του Ελσίνκη και με κάποια άλλα εργαλεία που διαθέτουμε μπορούμε να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και αυτή η σαφήνεια λέει ότι η εδαφική ακεραιότητα και η ελευθερία κάθε κράτους είναι αποκλειστικά και μόνο κυρίαρχη απόφασή του. Και το ε, κράτος θα πρέπει να μπορεί να αποφασίζει μόνο του για τις συμβάσεις και τις συνθήκες τις οποίες υπογράφει. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι επανερχόμεθα στις ε, κλασικές ε, πολιτικές, τις πολιτικές επίδειξης δύναμης του 19ου και του 20ου αιώνα. Αυτό λοιπόν αποτελεί ουσιαστική αλλαγή του σκηνικού. Δηλαδή για 25 ολόκληρα χρόνια θεωρούσαμε ότι όλες οι συγκρούσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΣΑ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, όπου εκεί γίνεται λόγος για την ε, μη διακριτική μεταχείριση των μειονοτήτων, για όλα αυτά εμείς πιστεύαμε ότι και οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ έχουν ρυθμιστεί. Κατόπιν τούτου θεωρούσαμε ότι γίνονται ειρηνικές και ήρεμες συζητήσεις. Δεν είναι έτσι όμως, αυτά αμφισβητούνται. Εν τω μεταξύ έχουν υπάρξει κάποιοι μηχανισμοί επίλυση διαφορών, όμως οι μηχανισμοί αυτοί αντικαθίστανται από την εξής θέση ότι όταν υπάρχουν ιστορικές διεκδικήσεις ή όταν δεν διαφυλάσσονται τα λεγόμενα εθνικά συμφέροντα, τότε δικαιούται κανείς να επανέλθει σε παλιές, σε υποτίθεται μη ισχύουσες πλέον αρχές, ότι μπορεί κανείς να λαμβάνει μόνος του τις δικές του αποφάσεις. Αυτό όμως είναι μία δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί αν ε, ισχύσει αυτό, τότε εγώ μπορώ να σου πω 100 θέματα για τα οποία θα μπορούσε να ξεσπάσει πόλεμο στην Ευρώπη, γιατί πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να πει έχω ιστορικές διεκδικήσεις και η εξελίξη στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δεν με ικανοποιούν. Στον 21ο αιώνα υποτίθεται ότι όλα αυτά τα έχουμε ε, ξεπεράσει, ότι έχουμε επιλέξει την ειρηνική συμβίωση. Δηλαδή υπάρχουν υποτίθεται στην Ευρώπη οι αρχές του διεθνούς δικαίου τις οποίες και σεβόμετα. Εάν όμως ε, αμφισβητούμε αυτές τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τότε τα πράγματα εξελίσσονται δυσάρεστα. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, ανεξάρτητα με την κριτική που ασκείται από τη Ρωσία, να καταφύγουμε σε στρατιωτικές επεμβάσεις. Ό,τι και αν γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές εφόσον τα πράγματα πήραν τις εξελίξεις που πήραν, ανεξάρτητα αν μας αρέσουν ή όχι, εφόσον λοιπόν διαπιστώνουμε ότι διεξάγεται πόλεμο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχει πόλεμος. Μία χώρα επιτέθηκε με στρατιωτικά μέσα σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό είναι πόλεμος. Νομίζω ο κύριος Σβάτσενπεχ το ανέφερε αυτό εχθές ε, στην παρέμβασή του. Αυτό λοιπόν το γεγονός σημαίνει ότι οφείλουμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική η οποία πρώτον θα ε, σκοπεύει στη διασφάλιση εγγυήσεων για τα ίδια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ είναι για άλλη μια φορά απολύτως απαραίτητο λόγω της συλλογικής ασφάλειας. Νομίζω αυτά τα είχαμε ξεχάσει. Ε, αυτό το είχε ξεχάσει και το ίδιο το ΝΑΤΟ. Σκεφτόμασταν το τι γίνεται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δεν σκεφτόμασταν όμως τι γίνεται με το ΝΑΤΟ. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όση κριτική και να ασκούμε απέναντι στις ΗΠΑ σχετικά με την ε, προστασία των δεδομένων και οτιδήποτε άλλο, αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε γιατί, γιατί εντάσσεται μέσα σε αυτή τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν όλα αυτά είναι θέμα συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι απολύτω σαφές ότι κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μακροπρόθεσμα πρέπει να έχει το ίδιο αίσθημα ασφαλείας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κράτη στην Ευρώπη τα οποία να βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα σε θέματα ασφαλείας. Νομίζω στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει αυτός ο θεσμός. Και αν συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη και η Ρωσία ε, συνεχίσει να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται με όλες αυτές τις ε, αεροπορικές ασκήσεις και τα παρεμφερή, τότε ενδέχεται κάποια στιγμή αυτό το χειμώνα να έρθει μια τέτοια χρονική στιγμή όπου το, ε, η συμφωνία του ΝΑΤΟ του 1997 με τη Ρωσία δεν θα ισχύει πλέον. Μέχρι τώρα, παρά προπαγανδιστικές δηλώσεις, η συμφωνία αυτή ισχύει. Και εκεί αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξουν δυνάμεις του ΝΑΤΟ ανατολικά του, Έλβα, του ποταμού Έλβα. Και αυτή η συμφωνία ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο συζητήθηκε στην Ουαλία είναι να υπάρξει η τήρηση αυτής της συμφωνίας και κάτω από αυτήν εκπεριτροπής ρυθμίσεις. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει γιατί όλα αυτά όπως σας είπα εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από τη συμπεριφορά της Μόσχας. Και πρέπει να σας πω ότι οι Πολωνία, οι Εστονοί, οι Λιθουανοί, Λετονοί, όλοι αυτοί οι φίλοι μας μου λένε, κοίταξε να δεις, εσύ ως Γερμανός οφείλεις να το καταλαβαίνεις αυτό περισσότερο από όλους διότι οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι στρατιώτες στο Δυτικό Βερολίνο και οι Καναδοί και όλοι οι άλλοι που βρέθηκαν στην Δυτική Γερμανία ήταν το όπλο σας. Αν υπήρχε τότε επίθεση των Ρώσων, αυτή θα ήταν η δική σας η ασπίδα. Είναι αυτοί που διασφάλιξαν διασφάλισαν την ειρήνη και στη τελική ανάλυση αυτή ήταν και η βάση για την ε, επανένωση των Γερμανιών. Και τώρα οι Πολωνοί φίλοι μου, ε, οι φίλοι μας, μας λένε με πόλη σαφήνεια, κοιτάξτε, επιθυμούμε και εμείς να απολαμβάνουμε την ίδια ασφάλεια, δηλαδή οι δυνάμεις αυτές να αποταλούν ε, όχι επιθετική, επιθετικό όπλο, αλλά να εγκατασταθούν για λόγους ασφαλείας. Ακριβώς όπως έγινε παλαιότερα και με τη Δυτική Γερμανία. Και πρέπει να σας πω ότι οποτεδήποτε μου το λένε αυτό, εγώ δεν βρίσκω κανένα αντεπιχείρημα. Και το ίδιο ισχύει οποτεδήποτε συζητάμε για την συνθήκη της Λισαβόνας και τη ρήτρα περί ε, παροχής ασφαλείας και βοήθειας. Ε, νομίζω λοιπόν ότι αυτό η στρατηγική φύση συζήτηση πρέπει να διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέλω που θέλω να πω είναι ότι κατά το επόμενο εξάμεινο θα προετοιμαστούμε ουσιαστικά και αυτό βέβαια θα γίνει και στα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί αυτό το θέμα θα αφορά κατά κύριο λόγο τις εθνικές κυβερνήσεις. Να προετοιμαστούμε λοιπόν για την συνάντηση κορυφής τον Ιούνιο, συνάντηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Πώς θα αντιδράσουμε λοιπόν. Όταν εμένετο ο ψυχρός πόλεμος ε, στην ε, Δυτική Γερμανία είχαμε 3.500 στρατιωτικά οχήματα που ήταν ε, αποτελεσματικό. έχουμε 250 που ούτε καν να τα χρησιμοποιήσουμε δεν μπορούμε. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εν τω μεταξύ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, στρατιωτικές ε, δυνάμεις ε, σε πολλά κρατημέλη με δαπάνες, ε, γενικές δαπάνες της τάξης του 78% που σημαίνει λειτουργεί με ένα μηχανισμός όμως δεν είναι αποτελεσματικές οι δυνάμεις αυτές. Στη Γερμανία μας είπανε αυτό δεν ισχύει, ε, οι συνολικές δαπάνες ε, ανέρχονται στο 48% είπα όμως ότι μια επιχείρηση που έχει συνολικές υπάγειες δαπάνες της τάξης του 48% θα πρέπει να κλείσει, είναι χροκοπημένη. Έχουμε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα, ε, η οποία υποτίθεται θα κάνει το συντονισμό στην έρευνα και την άμυνα. Εκεί εργάζονται 150 άτομα και Έχουμε και πολλές υπηρεσίες ε, στη Γερμανία που υποτίθεται ασχολούνται με αυτή τη διαχείριση των τεθωρακισμένων ε, και δεν μπορούν να προσφέρουν απολύτως τίποτα. Το ίδιο μπορώ να σας πω και για άλλα κράτη-μέλη. Για δέστε τώρα τη Γερμανία, 5.000 άνθρωποι, σαν να μην άλλαξε απολύτως τίποτα, με αποτελέσματα όμως που δείχνουν ότι τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη δαπανούν περίπου το 15% ε, για την άμυνα με αποτελεσματικότητα όμως 10%. Ξέρετε γιατί. Διότι δεν υπάρχει η αποτελεσματική συνέργεια, κάτι που χρειαζόμαστε. Υπάρχουν εδώ κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Α400M που είναι, ε, αυτό αφορά ένα πρόγραμμα μεταγωγικών αεροσκαφών. Σε τελική ανάλυση, δυστυχώς, και σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αεροπλάνα γιατί ήταν πολύ βαριά τα φορτηγά και πολύ αδύναμες οι μηχανές. Αυτό θα μπορούσε κανείς να το αντιγηθεί για ανέκδοτο, αλλά ξέρετε αυτό κόστησε ένα δισεκατομμύριο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και μπορώ να αναφέρω και πάρα πολλά άλλα παρεμφερή προγράμματα. Νομίζω, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ε, όσον αφορά την δυνατότητα άμυνας, είπαμε ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον εδαφική ικανότητα άμυνας. Λάθος ήταν αυτό. Λάθος που το είπαμε πριν από 5-6 χρόνια. Τώρα πλέον αυτή την ικανότητα άμυνας δεν μπορούμε να την επιτύχουμε με τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Οι Υπουργοί Άμυνας των κρατών μελών λένε δεν έχουμε πλέον τα απαραίτητα κονδύλια σε κανέναν εθνικό προπολισμό δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Και αν δω λοιπόν το τι πρέπει να κάνουμε με την κυβερνοασφάλεια σε όλες τις χώρες ε, έχουμε αναθέσει σε ερευνητές ε, να προβούν σε έρευνες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον ε, δεν υπάρχει καν κάποια εικόνα του ποιο κάνει τι. Ούτε και στο ΝΑΤΟ συμβαίνει αυτό. Έκανα πρόσφατα μία ομιλία και πραγματικά τρόμαξα. Όλοι δουλεύουν σε κάτι με κανέναν απολύτω συντονισμό. Καμία αποτελεσματικότητα αποτελεσματικότητα. Βεβαίως ε, και διότι όλα αυτά ε, πρέπει να ξέρουμε ότι συνδυάζονται και με βιομηχανικές απόψεις. Δηλαδή κάποιοι θέλουν να κερδίσουν και δεν θέλουν να κερδίσουν οι συναδελφοί τους. Ε, όμως το θέμα είναι ότι δεν μπορεί η βιομηχανική πολιτική να παρεμβαίνει στην κυβερνοασφάλεια η κυβερνοσφάλεια είναι καθοριστική σημασία γιατί είναι εκείνη που αποφασίζει σε περίπτωση πολέμου. Και αν δεν έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία, αν δεν έχουμε τους απαραίτητου κανονισμού, σίγουρα θα έχουμε προβλήματα. Όπως δεν μπορεί κανείς να ρυθμίσει και να ελέγχει το ίντερνετ σε εθνικό επίπεδο, ούτε και τον κυβερνοπόλεμο, το cyber warfare δεν μπορεί κανείς να ελέγξει. Γι' αυτό λοιπόν για μένα τίθεται το ερώτημα. Ε, σε επίπεδο έρευνας και συντονισμού, σε επίπεδο προμηθειών, δεν μπορούμε να λειτουργούμε από κοινού έτσι ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που κάνουν και οι Αμερικανοί με το 15%. Αυτή είναι η δραματική συζήτηση που θα λάβει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τους επόμενους μήνες. Και νομίζω ότι δυστυχώς με βίαιο και ομό τρόπο πρέπει να δούμε κατάματα την αλήθεια. Και πρέπει να το πράξουμε αυτό. Δεν ανέφερα και πολλά άλλα θέματα που υπάρχουν στην έκθεσή μου, αλλά σας τα είπα αυτά γιατί αυτά με απασχολούν ε, κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που μπορούμε να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. 11 ομιλητές ζήτησαν το λόγο και κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. Δύο λεπτά θα έχει ο καθένας για την ε, παρέμβασή του. Ας πούμε 1,5, 1,5 λεπτό. Ο καθένας ε, αγορητής θα έχει 1,5 λεπτό στη διάθεσή του. Ε, ακόμα ε, ας ανοίξουμε τον κατάλογο των μιλητών. Μπορείτε αν θέλετε να δηλώσετε και τώρα ότι επιθυμείτε το λόγο. Το λόγο έχει ο κύριος Κλίχ και μετά ο κύριος Πρέιντα. Κλίχ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έλμαρ. Σα ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μα έδωσε ε, να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Πολύ σωστά υπογράμμισε το ρόλο του θεσμικού πλαισίου για την κοινή πολιτική ασφάλειας και Άμυνα και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Και ευελπιστούμε ότι θα δημιουργηθεί μια νέα ηγετική τακτική και μια πιο ορθολογική χρήση των κονδυλίων. Πιστεύω ότι θα διδαχθούμε από το παρελθόν και θα επικεντρωθούμε στη συνοχή της ΚΕΠΑ. Θα είναι κλειδί την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Εγώ θα επικεντρωθώ στο τμήμα της έκθεσής σου που αφορά την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφυσβήτα έχουμε όλο και περισσότερες συγκρούσεις και κρίσεις και στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, κυρίως τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και την ε, ανάδειξη του Ισλαμικού κράτους. Δημιουργήσαμε ε, μία έξαρση των ε, εχθροπραξιών στην Ευρώπη και, ένα, και στη γειτονία της και ένα νέο κλίμα ασφάλειας που δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για το ΝΑΤΟ. Και θα πρέπει να προσδιορίσουμε τη φύση και το χαρακτήρα αυτών των κρίσεων. Σε ό,τι αφορά την ανατολική πλευρά της Ευρώπης, ε, ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να μετατρέψει τη Ρωσία από περιφερειακή δύναμη σε παγκόσμια δύναμη. Αυτή είναι η πρόθεσή του. Το θέμα είναι πού βρισκόμαστε εμείς και πώς θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και στη νέα απειλή που σίγουρα είναι η πιο δύσκολη γιατί είναι η πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου που έχουμε αναπροσδιορισμό των συνόρων στην Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον έχουμε δυστυχώς επιτυχής προσπάθειες υπονόμευσης του μοντέλου της διεθνούς ασφάλειας ενός μοντέλου που στηριζόταν μέχρι στιγμή σε διάλογο και συνεργασία και όχι στη χρήση βίας ή στρατιωτικής ισχύω. Αυτή τη στιγμή όμως ε, είμαστε μάρτυρες της κατάρρευσης αυτού του μοντέλου ασφάλειας που επικρατούσε τα τελευταία 20 χρόνια. Μέχρι στιγμής ε, δεν είχαμε επίθεση Ρωσίας ε, κατά χώρας ε, ΝΑΤΟ ή Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δημιουργούνται τόσες αναταραχές στα σύνορα που εύλογοι φόβοι προβληματίζουν τις χώρες μέλη και τους εταίρους μας ε, στο ΝΑΤΟ. Βραχυπρόθεσμα πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση των ε, όρων και προϋποθέσεων της Συμφωνίας του Μίνσκ. Γιατί παρά την υποχρεωτική εκεχηρία η κατάσταση είναι αβέβαιη. Βέβαια αυτή η τακτική της Ρωσίας είναι γνωστή, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις πιέσεις για να επανέλθουμε στην τήρηση της Συμφωνίας Μίνσκ. Και πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα πρέπει να επιστρέψουμε στην παλιά μορφή και μοντέλο συνεργασίας και να κρατήσουμε αμύωτη την πίεση προς τη Ρωσία για να επανέλθει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν κύριε Πρόεδρε να σας συγχαρώ για το έγγραφο εργασίας σας που από των βασικών θεμάτων της κοινή πολιτικής ε, εξωτερικών ασφάλειας και άμυνας και δίνει προτεραιότητα στην ε, ανάγκη διαμόρφωσης μιας στρατηγικής προσέγγισης στην ε, εξωτερική μας πολιτική. Χθες ακούσαμε κάποιο δεικτικό χρονοδιάγραμμα από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και ελπίζω να επανέλθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ξανασυζητήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους στρατηγικούς μας εταίρους. Και κάτι τέτοιο επίγει, γιατί έχουμε και την συζήτηση και το θέμα της Ρωσίας. Γιατί όπως λέτε στην παράγραφο 20, θα πρέπει να καλέσουμε τη Ρωσία σε έναν αξιόπιστο διάλογο και επίσης να λάβουμε υπόψη την πράξη του Ελσίνκη του 1975, γιατί είναι σαφές ότι σήμερα η Ρωσία δεν εστερνίζεται τις ίδιες αρχές και αξίες με εμάς. Και παραβιάζει και την συμφωνία του Ελσίνκη του 1975. Και για τα δημοσιονομικά θέματα έχετε δίκιο, γιατί θα πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, να εφοδιαστούμε με τα κατάλληλα μέσα και τη σωστή χρηματοδότηση. Και επίσης θέλουμε μια ταχύτερη διαδικασία για να μπορούμε να αντιδρούμε πιο άμεσα στις κρίσεις που ανακύπτουν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Good morning. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Θα ήθελα Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δίνεται να λάβουμε μέρος στη συζήτηση και συγχαρητήρια στον Έλμαρ Μπροκ που κάλεσε τους Προέδρους των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εστερνίζομαι και εγώ την ιδέα ότι από την 1η Δεκεμβρίου έχουμε μια ολοκένουργια Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια νέα κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και μια νέα κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άποψη αυτή. Και επίσης θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια τελείως νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας. Το 2003 είχαμε την τελευταία συμφωνία για την πολιτική ασφάλεια, τώρα χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία όχι ανανέωση της παλιάς, γιατί δημιουργείται πια ένα νέο πλαίσιο και περιβάλλον ασφάλειας. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες ε, και τα χαρακτηριστικά αυτού του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας, γιατί μας, ε, ανέπτυξε, μας τα ανέπτυξε εκτενώς ο Έλμαρ Μπλοκ. Εγώ θα επικεντρωθώ σε ένα σημείο. Ναι, όντως η Ρωσία φαίνεται ότι επανέρχεται στις επεκτατικές και αυτοκρατορικές, αυτοκρατορικές της τάσεις. Θα πρέπει να πούμε όχι σε αυτή την πολιτική δημιουργία σφαιρών επιρροής και λέμε όχι στην επαναφορά της εποχής του ψυχρού πολέμου και στο διχασμό της Ευρώπης με τύχη. Πιστεύω πάντως ότι όταν διαμορφώσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική και στρατηγική ασφάλειας είναι σημαντικός ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί πια έχουμε πολύ καλύτερη ευκαιρία για ενισχυμένη συνεργασία στο μέλλον δεδομένων και των νέων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς τα εθνικά κοινοβούλια συνεχώς αναζητούμε τον κοινοβουλευτικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, γιατί δεν καθοδηγούμε εμείς την ε, εξωτερική πολιτική σε καθημερινή βάση, αλλά συμβάλλουμε στη δημιουργία στρατηγικών ε, και για κάτι τέτοιο χρειάζεται μια ευρεία πολιτική συνένεση με συμμετοχή της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό θα είναι αποφασιστικός ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση ε, των διαφόρων στρατηγικών συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή τη συζήτηση, λέει η κυρία Γκόμες. Πράγματι πρέπει να ξαναδούμε την ε, πολιτική μας αυτή, την κοινή εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλεια εξαιτία της Ρωσίας. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη δράση της Ρωσίας πολιτικά, πρέπει να έχουμε και του στρατιωτικού μυς που μα χρειάζονται για να κερδίσουμε σε αξιοπιστία. Και στηρίζω βέβαια την αναθεώρηση της στρατηγικής μας, της ευρωπαϊκής. Συγχρόνως όμως πρέπει να επικεντρωθούμε και στα αποτελέσματα της ήδη υπάρχουσας πολιτική μας. Γιατί αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία, έχει να κάνει με το ότι δεν είχαμε προετοιμαστεί όντω καλά υπό την τρέχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική. Συνεπώς πρέπει να εξαναδούμε το δημοσιονομικό ζήτημα του προπολογισμού, μια κοινή χρηματοδότηση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι ζωτική σημασίας. Και το έχουμε ζητήσει ξανά και ξανά. Πρέπει επίσης να προσέξουμε πολύ το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Χρειάζεται βέβαια πολιτική βούληση και αυτό έλειπε μέχρι τώρα και είναι κρίμα που δεν είχαμε τέτοιου είδου ηγετικό ρόλο από πλευράς της Lady Άστον. Ε, θα μπορούσε, αλλά δεν το έκανε. Και βέβαια, συνεπώς δεν μπόρεσε να κερδίσει και τις χώρες μέλη. Κάτω από τις συνθήκες της κρίσης, μάλιστα, τα πράγματα χειροτέρεψαν και τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, που βέβαια ήταν και αυτό θέμα πολιτικής βούλησης, τελικά καταλήξαμε να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει για να προετοιμαστούμε καλά στον τομέα της ασφάλειας. Ουσιαστικά καταστρέψαμε τις ικανότητες που είχαν κάποιες χώρες όπως η δικιά μου. Μάλιστα θα έλεγα ότι ξεπουλήσαμε και πολύ σημαντικούς τεχνολογικούς τομείς στον τομέα της ασφάλειας και της άμενας, στους Κινέζους και σε άλλους. Θα το πληρώσουμε αυτό ακριβά. Και αν δεν αλλάξει αυτό πολύ γρήγορα θα χειροτερέψει η κατάσταση ακόμα περισσότερο. Ένα λεπτό καθένας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, μην καθυστερείτε πολύ. Ο κύριος Καζίνη. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Τρία πράγματα θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ ότι η Επιτροπή εδώ, τις οποίες προείσταστε, θα πρέπει να ε, βοηθήσει στο συντονισμό ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβουλία. Περισσότερο στο μέλλον. Γιατί δεν θα υπάρχει εξωτερική πολιτική και ε, πολιτική κοινή άμυνα αν δεν υπάρχει και καλύτερο συντονισμός ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια. Επ' αυτού λοιπόν, το να βλέπει κανείς σήμερα το πρωί στην ε, τηλεόραση, στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα ότι το Γαλλικό Κοινοβούλιο σχετικά ε, με το θέμα της αναγνώρισης ε, της ε, Παλαιστίνης γίνονται συγκεκριμένες συζητήσεις, αυτό πρέπει να σας πω ότι εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί δεν μπορούμε έτσι να έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Δεν είμαστε αξιόπιστοι όταν βλέπουμε ότι οι Μογκερίνοι και άλλοι προβαίνουν σε μια κοινή εξωτερική πολιτική και οι υπόλοιποι δεν ακολουθούν μια τόσο εμβληματική απόφαση όπως είναι η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Προφανώς και είναι συμβολική όλη αυτή η συζήτηση. Οι κυβερνήσεις είναι εκείνες που δίνουν εντολή στα κοινοβουλία, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη ευκαιρία για να δείξουν τα κοινοβούλια ότι είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν με μια κοινή εξωτερική πολιτική. Η δική σας η Επιτροπή, της οποίας αναγνωρίζουμε τον ηγετικό ρόλο, θεωρώ ότι μπορεί να παίξει συντονιστικό ρόλο ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια. Ε, οι δικές μας εξωτερικές επιτροπές, τουλάχιστον της Γερουσίας, Λευκορωσίας και του δικού μα του Κοινοβουλίου στην Ιταλία είναι ε, πρόθυμες να σας βοηθήσουν. Πάμε τώρα στη Ρωσία. Στην ε, Ιταλία λέμε ότι οι καλύτερες προθέσεις οδηγούν μέσα από την κόλαση. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε γιατί αυτά τα οποία έγιναν τους τελευταίους μήνες, να λέμε παραδείγματο χάρη, ότι η Ουκρανία πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ, αυτό σημαίνει ότι διαδίδονται και μεταφέρονται αυταπάτες γιατί η Ουκρανία δεν μπορεί να μπει στην Ευρώπη. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ουκρανία και η αλληλεγγύη προς την Ουκρανία είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να εξτάσουμε όλοι από κοινού αλλά αυτή η αλληλεγγύη, για να είμαστε ειλικρινεί, έχει ένα συγκεκριμένο κόστος. Το να κατεβαίνει κανείς στους δρόμους και να λέει δείχνουμε αλληλεγγύη προς την Ουκρανία, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη. Γιατί αλλιώς αυτά τα οποία λέμε είναι απλώς μεγαλοστομίες. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Thank you very much, Chairman. Well, um, I Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Φανόρδεν. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η ανάλυση σας για όλα αυτά τα χρόνια ήταν στραβή. Η απάντηση για σας είναι περισσότερη Ευρώπη. Αυτό ζητάτε, περισσότερη Ευρώπη. Και έχουμε ανακαλύψει εκ νέου το ΝΑΤΟ. Όμως η ιστορία και η εμπειρία θα έπρεπε να μας διδάξει ότι η Ένωση των Δημοκρατιών είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Έχουμε μια ισχυρή οργάνωση και αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Ενώ τι κάνουμε εδώ, είναι ότι κάνουμε μια γελία παντομήμα προσπαθώντας να φτιάξουμε αυτόνομες δομές παράλληλα με το ΝΑΤΟ όπου συμμετέχουν λίγο πολύ ίδιες χώρες καταστρέφοντας έτσι πολιτικά το ΝΑΤΟ και κατασπαλώντας ε, πόρους. Είναι τρελό. Θέλετε τα ίδια να ισχύουν για την άμυνα όσα προβλέψατε και για το ευρώ. Όλα αυτά τα αρνητικά. Και με τι στόχο, επειδή συνεχίζεται αυτό το όνειρο, αν θέλετε να το πω έτσι, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ενώ θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στην άμυνα και την ασφάλεια των εθνών μας. Πρέπει να δώσουμε νέα πνοή στο ΝΑΤΟ, να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και χρειάζεται σίγουρα πολιτική βούληση. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να σταματήσουμε να στρεφόμαστε αλλού αντί να επικεντρωνόμαστε σε αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να το πάρουν πίσω στις χώρες τους τα εθνικά κοινοβούλια. Αλλά βέβαια δεν συμφωνούν ε, όλοι, πρέπει να ξέρετε, με την ιδέα αυτή ότι η λύση για οποιαδήποτε κρίση και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα είναι η περισσότερη Ευρώπη. Τζόφρι, νομίζω με παρεξήγηση δεν με κατάλαβες καλά. Ε, εγώ είπα ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ολοκλήρωση για να μπο... είμαστε σε θέση να αναπτύσσουμε ικανότητα, στρατιωτική ικανότητα που ε, θα είναι αποτελεσματική μέσα στον ΝΑΤΟ η Ενωμένη Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει το ΝΑΤΟ, να είναι το ΝΑΤΟ ισχυρό. Νομίζω ότι μέχρι και σήμερα δεν το έχεις καταλάβει αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν θες να το καταλάβεις. Ε, Έλμα, ε, εγώ θα προσπαθήσω αυτά που είπες ε, να τα δω κάτω από καλή σκοπιά. Ναι, λέει ο κύριος Μπρόκ, αλλά θα πρέπει αυτά που είπα να τα εξετάσεις στο σύνολό τους και όχι αποσπασματικά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και θα πρέπει να τεθεί προσυζήτηση και στο Συμβούλιο. Ήδη είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανίκανη ε, να αντιδράσει άμεσα και να δώσει αποτελεσματικές λύσεις ε, σε σημαντικές κρίσεις ε, με δραματικές συνέπειες, όπως αυτές που είχαμε στην Ευρώπη και στη γειτονία της. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνοχή, τη δράση και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική πολιτική. Αυτό βέβαια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από το Συμβούλιο και από τα κράτη-μέλη, αλλά και από την επιρροή που θα ασκήσουν στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρώπη είχαμε μια ανησυχητική έξαρση αντιευρωπαϊκών και λαϊκιστικών δυνάμεων που μακροπρόθεσμα μπορούν να υπονομεύσουν και το ευρωπαϊκό όραμα και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Και ήταν ανίκανη η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώ να αντιδράσει. Για παράδειγμα, στην κρίση ε, με τη Ρωσία δεν ε, δημιουργήσαμε, δεν διαμορφώσαμε ένα στρατηγικό όραμα για να αντιμετωπίσουμε την, ε, τον πόλεμο στην Ουκρανία ή την αποτυχία σύναψη συμφωνιών με τις χώρες της πολιτικής γειτονίας. Επίσης αποτύχαμε στην διαχείριση της μετανάστευσης στη Μεσόγειο ούτε καταφέραμε να στηρίξουμε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου κράτους στην Παλαιστίνη, εξαιτίας της έλλειψης συντονισμένης και αποτελεσματικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ερωτώ λοιπόν και γιατί αυτή η ανικανότητα. Πιστεύω ότι για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να αλλάξουμε τις διαρθρώσεις μας και τον τρόπο δράσης μας. Θέλουμε πιο συντονισμένη εξωτερική δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με περισσότερα κράτη-μέλη που θα συμμετέχουν σε αυτή. Είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο διαρωτώμα. Ευχαριστώ. Κύριος Αουστρεβίτσιος. Um, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει. Βλέπουμε ανατολικά έναν υβριδικό πόλεμο, ο οποίος απαιτεί υβριδικές απαντήσεις. Κάτι διαφορετικό από ό,τι κάναμε κατά το παρελθόν. Πρέπει να αντιληφθούμε διαφορετικούς κινδύνους κάτω από τη διαφορετική μορφή όπου φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, το θέμα του κυβερνοχώρου και της ενέργειας και ασφάλεια σε αυτά χρειάζονται αποτελεσματική και έγκαιρη απάντηση μέσω της ενημέρωσης. Προς το παρόν το χάνουμε αυτό το πόλεμο. Έχουμε συνεχώς επίθεση με προπαγάνδα. Οι ευρωπαϊκές αξίες και η ευρωπαϊκή πολιτική επικρίνονται συνεχώς. Και αν νομίζουμε ότι η τιμή της αλληλεγγύης προς την Ουκρανία είναι υψηλή, η τιμή της μη αλληλεγγύης θα είναι ακόμα υψηλότερη. Το λόγο έχει κυρία Ιντότερο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Είμαι από τη Ρουμανία, από τη Ρουμανική Βουλή και θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Μπρόκ για την ε, εμπεριστατωμένη έκθεσή σας ε, για την κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Θα αναφερθώ στην παράγραφο 21 της έκθεσής σας. Δεδομένη στις θέσεις της Ρουμανίας ε, για την Ανατολική Γειτονία και ιδιαίτερα τη θέση μας απέναντι στην Μολδαβία, θεωρώ ότι η σύναψη συμφωνία σύνθεσης με τη χώρα αυτή είναι σημαντική. Χώρες όπως η Μολδαβία σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην ενταξιακή τους προοπτική και αυτό θα πρέπει να τις στηρίξουμε. Χαιρόμαστε για τα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης στη Μολδαβία. Έδειξαν ότι ο λαός της Μολδαβίας έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι γι' αυτό και η Μολδαβία χρήζει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση με όλο και περισσότερα βήματα. Η κυρία Λόιζον, που είμαι σίγουρη, σίγουρος ότι θα με υπερασπιστεί σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Βανόρντεν. Προφανώς και θα το κάνω, και επίσης ε, χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση. Θέλω όμως να πω ότι το 1,5 λεπτό που μας δώσατε είναι πολύ λίγος χρόνος, κυρίως όταν πρόκειται για πολύ ειδικά θέματα, όπως ε, θέματα που αφορούν στον έλεγχο των ε, προϋπολογισμών. δεν μπορεί κανείς να αναφερθεί σε όλα αυτά, γι' αυτό και εγώ θα περιστώ σε κάποιες γενικής φύσεως παρατηρήσεις. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι χαίρομαι για την έκθεση του Πρόεδρου τη βρίσκω πάρα πολύ καλή, βρίσκω πολυθετικό το πόσο ο πρόεδρος ε, παρουσίασε με απόλυτη σαφήνεια τις κατευθυντήριες γραμμές της εξωτερικής πολιτικής. Ε, και πρέπει να σας πω ότι με απόλυτη σαφήνεια καθίσταται σαφές ε, ποιες είναι οι αρχές που πρέπει να ισχύουν στην έκθεση και σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος κατέστη απολύτως σαφές το ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιος παίκτη. Βέβαια πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει παγκόσμιος παίκτη. Για μας παγκόσμιος παίκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει περισσότερη δύναμη και επιρροή. Και όπως είπε ο κύριος Μπροκ, εδώ Πρόκειται για την ελευθερία των επιχειρήσεων, των πολιτών, κάτι που δυστυχώς δεν το σκεφτόμαστε συχνά. Αυτό που ενδιαφέρει είναι κυρίως μεγαλύτερη εξουσία, μεγαλύτερη επιρροή, ε, Υποτίθεται γίνονται κάποιες αναφορές σε ανθρωπιστικές ιδέες της ε, Ευρώπης ε, που πρέπει να εφαρμόζονται στον υπόλοιπο τον κόσμο. Χρησιμοποιούνται όμως ε, και στρατιωτικές δυνάμεις για να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξουσία και μεγαλύτερη επιρροή και οποτεδήποτε αποτυγχάνει αυτό το εγχείρημα τότε διρωτώνται μερικοί μήπως ήταν λάθος από τη σύλληψή του. Προχωράει η στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό ισχύει και με τον Πούτιν και χαίρομαι που μόνο σε μένα πάντα προσέχετε πόσο χρόνο μίλησα. Όχι, λέει ο πρόεδρο, ξεπεράσατε το χρόνο που σα διέθεσα κατά 50 δευτερόλεπτα. Άρα βλέπετε ότι ήμουν ιδιαίτερα γενναιόδωρο απέναντί σα και παρεπιπτόντω Εγώ δεν μίλησα ε, για την ελευθερία των επιχειρήσεων και των πολιτών να ανατρέξετε παρακαλώ στο κείμενό μου και να το διαβάσετε. Το λόγο έχει τώρα ο Fürst von Schwarzenberg. Ο κύριος Μπροκ ε, πολύ σωστά επισήμανε ότι όλοι οι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα στην ίδια ασφάλεια. Μόνο που σε κάθε χώρα υπάρχουν κάποιες περιοχές ε, της χώρας που δεν νιώθουν ίδια ασφάλεια. Ε, βλέπουμε να δραστηριοποιούνται συμμορίες και παρεμφερεί. Εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ έχουμε δηλώσει ότι εκεί όπου είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος Καλύτερα να υπάρχουν λιγότεροι αστυνομική γιατί ενδέχεται αυτό να αποτελεί πρόκληση και για τους βιαστές και για τους ληστές. Ε, και γι' αυτό θεωρούμε ότι εκεί που υπάρχει κίνδυνος καλύτερα να υπάρχουν και λιγότερες στρατιωτικές δυνάμεις. Αν δω μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τι συμβαίνει με το στρατό, εγώ ε, σας συστήνω να δείτε λιγάκι στην τηλεόραση, τηλεοπτικές ε, καταγραφές για το τι συνέβη στην Ουκρανία και στην ε, Κρυμαία με την ρωσική εισβολή. Ποτέ δεν έχω δει τόσο σύγχρονη τεχνολογία στη σημερινή εποχή, άριστη κατάσταση των τεθωρακισμένων, άριστη η επικοινωνία των στρατιωτών μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Καμία σχέση με τη στρατιωτική μηχανή της Σοβιετικής Ένωσης του προηγούμενου αιώνα. Thank you, Chair. I might not even need my 90 seconds for... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν χρειάζομαι καν τα 90 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε και μάλιστα με τα εθνικά κοινοβούλια. Πιστεύω εμείς οι πράσινοι συμφωνούμε με το τελευταίο κομμάτι για τη νέα τάξη πραγμάτων, αλλά θέλω να διευκρινίσω ένα ζήτημα. Παρακαλώ, στην παράγραφο 21 μιλάμε για την ανατολική εταιρική σχέση. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη δέσμευση για την διαδικασία σύνδεσης στην περιοχή. Πρέπει όμως να ξαναδούμε το ρόλο γενικότερα της ανατολικής αυτής ε, εταιρικής σχέσης στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής ασφάλειας. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Ευχαριστώ, Έλμαρ. Η κυρία Μογκερίνη χτες είπε δύο φορές ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τη Ρωσία. Η δικιά μου απάντηση είναι ότι έχουμε στρατηγική για τη Ρωσία και ότι η στρατηγική αυτή λειτουργεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσουμε ειλικρινά και απόλυτα τίμια ότι οι δυνατότητες πολιτικού διαλόγου με την Ρωσία έχουν εξαντληθεί και ότι πρέπει να συνεχίσουμε με την δικιά μας στάση υπέρ κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εάν η Ρωσία λάβει συγκεκριμένα βήματα να φύγει από την Ουκρανία, τότε μπορεί να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα ένα κόσμο όπου η ευρωπαϊκή προοπτική, η ενταξιακή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια δεν θα είναι κάτι που θα αναφέρεται μόνο στα ψηφίσματα και στα χαρτιά, αλλά μία εφικτή προοπτική. Τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα της στρατηγικής μας. Ακόμη και αν η διεύρυνση έχει προς το παρόν ε, διακοπή και από ό,τι ακούσαμε δεν αναμένεται νέα διεύρυνση την επόμενη πενταετία. Οτιδήποτε άλλο όμως θα ήταν εσφαλμένο. Θα πρέπει να απεμπλέξουμε αυτή τη διαδικασία, να την απελευθερώσουμε. Γιατί υπάρχουν κίνδυνοι στη Βοσνία Ερσεγοβίνη, στη Μακεδονία για παράδειγμα, λέει ο μιλητής. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε την ενταξιακή διαδικασία αυτών των χωρών, γιατί άλλες χώρες ε, θα προσπαθήσουν να τις προσελκύσουν. Ε, θα πρέπει να έχουμε συνέργεια στους, ε, στα θεσμικά μας όργανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβουλία. Πολύ σημαντική η συνεργασία αυτή, κυρίως διότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ απαραίτητο να βαδίσουμε μαζί. Ε, την κρίση στην Ουκρανία-Ρωσία δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως ε, περιφερειακή κρίση γιατί αν ήταν έτσι θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε με τη συμφωνία της Βουδαπέστης και εγώ διερωτώ με γιατί δεν το έχει σκεφτεί κανείς ποτέ μέχρι σήμερα αυτό η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία επιθυμεί να επαναφέρει το δόγμα του Μπρέζνεφ του 86 ότι τα σύνορα των κρατών κρίνονται και ανάλογα με τα σοσιαλιστικά συμφέροντα. Αυτό ελέγχθη κάπως και εδώ χθες. Ε, αυτό που με ξενίζει είναι ότι, εντάξει, ακούστηκαν πάρα πολλές ε, λεπτομέρειες, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίσουμε συμπαγός αυτή την επιθετικότητα που δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά την ευρωπαϊκή κοινότητα αξιών. Ευχαριστώ κύριος Πάσκος και όδησε εισηγητής είναι ομιλητής και μου ζήτησε να, σε μια άλλη εκδήλωση και μου ζήτησε να παρουσιάσω τις θέσεις του. Θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το έγγραφο εργασία, το οποίο μας προσφέρει μια βάση για να συζητήσουμε τα θέματα κλειδί. Το έγγραφο εργασία είναι καλά επεξεργασμένο και μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι θα συνεχιστεί η ίδια δομή η οποία θα επικεντρώνεται σε νέες συστάσεις με περιφερειακή προσέγγιση για τα θέματα κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλεια. Πιστεύω, κύριο Πάσκου, ότι θα πρέπει να είναι πιο δυνατή. Υπάρχουν δύο επιχειρήματα για πιο ισχυρέ κατευθυντήριε γραμμέ στην έκθεση αυτή. Αφενό, πρόκειται για την διαφορά στο περιβάλλον που υπάρχει τώρα στην ε, στις χώρε που βρίσκονται ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δεύτερο λόγος είναι ότι έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νέα ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται περισσότερη συνεχή στη, συνοχή στην εξωτερική μας πολιτική ασφάλειας και προτάσεις οι οποίες να μας ε, οδηγούν στο στόχο μας αυτό. Επίση, πρέπει να υπάρξει νέα πολιτική στρατηγική, καλά διαρθρωμένη, που να δημιουργεί μια νέα τάξη. Πράγματα τα οποία αναφέρονται και στην τελική πράξη του Ελσίνκη και δεσμεύει όλε τι χώρε μέλη συμπεριλαμβανομένη και τη Ρωσία. Συμφωνεί κύριο Πάσκου πάντω για τι τις προτεραιότητε τη πολιτική μα αυτή για έλεγχο, σταθεροποίηση στην, ε, στις χώρες ανατολικά της Ευρώπης. Και συμφωνεί με το πνεύμα αυτό. Συμφωνεί επίση ότι η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να βασίζεται σε θέματα τα οποία είναι προ το συμφέρον ολόκληρη τη Ευρώπης και να βασιζόμαστε σε μια κοινή αντίληψη για το τι επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Υπάρχουν και άλλα σημεία βέβαια, αλλά με περιορίζει ο χρόνο, δεν θα πω τίποτα άλλο, αλλά θα σα τα υποβάλω αργότερα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ θέλω να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή. Ο Επίτροπος αν είπε χτες ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα των ε, γειτόνων μας. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με την παγκοσμιοποίηση και έχουμε να κάνουμε μια νέα τάξη στον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ότι χρειάζεται μια νέα στρατηγική ασφάλειας, πιστεύω, και σχέσεων με τον ΝΑΤΟ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αναλύσουμε κατά πόσο οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη βρίσκονται στον ίδιο δρόμο και στηρίζουν τα ίδια συμφέροντα. Μερικέ φορέ υπάρχουν διαφορετικά γεωπολιτικά συμφέροντα ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα στη δικιά μα πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε τη όσον αφορά την άμυνα αλλά το να δώσουν περισσότερα χρήματα οι χώρες μέλη χωρίς να υπάρχει τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα είναι πεταμένα χρήματα κατά τη γνώμη μου. Πρέπει λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες να δούνε τι θα γίνει και με την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων. Η ευρωπαϊκή σταθερότητα πάντως και η ασφάλεια απαιτεί και νέα πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Είχαμε μια καλή στρατηγική απέναντι στη Ρωσία και πρέπει να δούμε κατά πόσο σε αυτήν την Ήπειρο θέλουμε ασφάλεια διαρκείας και σταθερότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα έπρεπε να σας το έχω πει ότι μιλάμε για τη διαρθρωτική συνεργασία για συνεργασία σε θελοντική βάση. Αυτό ίσως όντω είναι ένα κομμάτι που πρέπει να ενισχύσω περισσότερο στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω πολωνικά για να δουλέψουν και οι διερμηνείς ε, από τα πολωνικά. Εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση, οποιασδήποτε επιτυχίες της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και της κοινή πολιτικής άμυνας ε, είναι η διαρθρωτική συνεργασία και η κοινή αντίληψη των ε, απειλών και των προκλήσεων. Και με αυτή την κοινή αντίληψη είχαμε τα τελευταία χρόνια πρόβλημα. Επιπλέον, ε, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε συνεννόηση για τα θέματα αυτά και κοινή αντίληψη, έχουμε και τη σημερινή κατάσταση ε, με τη Ρωσία. Και σε κάποιο βαθμό Έχουμε πρόβλημα και στο Ιράκ και τις απειλές από το αποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος, το ΙΣΙΣ. Αυτά μας είπε προηγουμένως και ο πρόεδρος. Μερικές φορές αντιμετωπίζουμε κάποιες ε, ε, σχέσεις μας ε, υπό, το, υπό την εμπορική σκοπιά ή σαν να μην συμβαίνει τίποτα ιδιαίτερο. Ίσως αυτό ήταν αφέλεια δική μας ή δεν δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιες προκλήσεις. Επίσης, όταν εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δεν ενημερώθηκαν ε, για τίποτα ουσιαστικά δεν είπαν ότι δεν θα, έχουμε καμία δραστηριότητα του ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να, να εμείνουμε στην αρχή της αλληλεγγύης και στην κοινή αντίληψη, της συνεννόηση μεταξύ των συμμάχων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Νομίζω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Θεμελιώδες θέμα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν έχουμε χρόνο, ούτε έχουμε την πολυτέλεια της επικάλυψης των προσπαθειών. Γι' αυτό προτιμώ τις δράσεις να τις αναλάβουμε σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Δυστυχώ πρέπει να σταματήσουμε τώρα συζήτηση, γιατί έτσι κι αλλιώ εδώ και ένα τέτοιο θα περιμένουν έξω από την πόρτα οι έξι Υπουργοί Εξωτερικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτέ τι ε, παρεμβάσει σα και θα ήθελα ε, να προσκαλέσω τόσο εσάς όσο και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων κατά τις αμέσως επόμενες εβδομάδες να μου καταθέσετε προτάσεις, ε, βελτίωσης γιατί προτίθεμαι να ε, συντάξω την έκθεσή μου πριν από τα Χριστούγεννα. Και τέλη Ιανουαρίου ε, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Πολύ βέβαια εξέφρασαν απόψεις ε, που στηρίζουν ε, τις θέσεις μου και αυτά θα τα συμπεριλάβω στην έκθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τη συζήτηση. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τους ε, Υπουργούς Εξωτερικών. Η διαδικασία θα είναι η εξής. Θα μιλήσουν με αλφαβητική σειρά οι Υπουργοί Εξωτερικών. Μετά θα λάβει το λόγο ο εισηγητής μας για κάθε μία χώρα και μετά θα ξεκινήσει η ευρύτερη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η βέλτιστη οργάνωση της συνάντησής μας. Σας ευχαριστώ πολύ.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 να καλωσορίσω τους ε, Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να διευκρινίσω ότι η Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι υπέρ της Συμφωνίας της Θεσσαλονίκης, εμένη στη Συμφωνία της Θεσσαλονίκης δηλαδή στην πρόσκληση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να γίνουν μια μέρα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν έχουμε κανένα λόγο να απομακρυνθούμε από την πολιτική αυτή. Και αυτό που συζητούμε τελευταία πέντε χρόνια είναι τεχνικά θέματα που δεν προϋποθέτουν καμία καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι σαφές από μας. Και μάλιστα χθες ο Επίτροπος Χάν και η Πατεκπρόσωπος Μογκερίνη δήλωσαν ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Θεωρούμε ότι οι χώρες αυτές ανήκουν στην Ευρώπη και αν θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τους περιμένουμε με ανοιχτέ αγκάλες γιατί θεωρούμε ότι η ένταξη αυτή είναι προς το αμοιβαίο μας συμφέρον. Θα σας βοηθήσουμε λοιπόν και πολιτικά και διπλωματικά και οικονομικά και όπως μπορούμε με κάθε τρόπο για να υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα και να βρούμε λύση με κάθε τρόπο. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον Ράμπο Κουβοκάβιτς, τον πρόεδρο της Βουλής του Μαυροβουνίου. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Θα δώσω τώρα το λόγο πρώτα στους Υπουργούς Εξωτερικών το λόγο με τη αλφαβητική σειρά των χωρών τους. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, τον κύριο Μπουσάτια. Thank you. Ευχαριστώ. Για πέντε λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπροκ, λέει ο κύριος Μπουσάτη. Επιτρέψτε μου να αρχίσω τις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις εκφράζοντας σας την ευγνωμοσύνη μου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους Ευρωβουλευτές που με συνέπεια στηρίζουν τη διαδικασία προσχώρησής μας και στηρίζουν γενικότερα την διαδικασία προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλω να σας πω δύο λόγια για τη διαδικασία προσχώρησης της Αλβανίας. Τον Ιούνιο που μας πέρασε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να δώσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Αλβανία. Η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέτος υπογραμμίζει την πολιτική βούληση των αρχών της Αλβανίας και της κυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά την διαδικασία αυτή. Εμείς βλέπουμε έτσι καλλιώς σαν προσωρινό βήμα το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε με μια αξιόπιστη διαδικασία με προβλεπόμενη ημερομηνία για την προσχώρησή μας και θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν κυρίως στην οικονομία και στο κράτος δικαίου καθορίζοντας κριτήρια για τα κεφάλαια 23 και 24. Για να πετύχει η διαδικασία ένταξη σίγουρα πρέπει να είναι δυναμική και αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν χαιρόμαστε πολύ που έχει υπάρξει οικονομική διακυβέρνηση σαν βασικός πυλώνας της διαδικασίας αυτής. Φέτος η Παγκόσμια Τράπεζα έβαλε στη δεσακοστή θέση την Αλβανία εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων της στην οικονομία και το κράτος δικαίου. Συνεπώς, η οικονομική διαδικασία αποτελεί ακρογωνία ολίθο για την διαδικασία μας. Προχωρούμε επίσης και στην οικοδόμηση του κράτους με νομοθεσία για την συμμόρφωση προς τον νόμων προκειμένου να καταστρέψουμε εγκληματικούς παραδείσους και να προχωρήσουμε σε θέματα όπως είναι η ενέργεια, που είναι ένας από τους βασικούς τομείς, και την αξιοπιστία του προϋπολογισμού με πάνω από 150 εκατομμύρια. Επίσης αυτό που κάνει η Αλβανία είναι προχωράει και σε άλλες δομές νομικές, πράγματα τα οποία εμείς ονομάζουμε με τον γενικό τίτλο «Οικοδόμηση δικαίου στη χώρα». Έχουμε πέντε προτεραιότητες προκειμένου να αρχίσουν οι συνομιλίες. Για μας η πιο σημαντική προτεραιότητα είναι η μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και οι μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, που αποτελεί σίγουρα ε, κάτι που βοηθάει την περιφερειακή ολοκλήρωση, γιατί δημιουργεί υγιή ανταγωνισμό στην περιοχή. Ο δεύτερος τομέας είναι η περιφερειακή συνεργασία. Τους τελευταίους μήνες είδαμε έντονη δράση σε αυτόν τον τομέα. Γίνεται πολλή δουλειά στα Δυτικά Βαλκόνια. Προσπαθούμε να είμαστε μια περιφέρεια και πολιτική και οικονομική. Η κρίση βέβαια στην Ουκρανία έδειξε ότι πολιτικά υπάρχουν δυσκολίες, διότι οι χώρες αντέδρασαν διαφορετικά στην κρίση καθεμία. Οικονομικά Ακόμα δεν είμαστε μια περιφέρεια γιατί δεν υπάρχει αρκετή σύνδεση. Και όσον αφορά την ασφάλεια, ούτε και εκεί ακόμα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μια περιφέρεια. Προσπαθούμε λοιπόν να μπούμε σε νέες πολιτικές σχέσεις στην περιοχή. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργό μας Ράμα πήγε στη Σερβία και αυτό αποτέλεσε κάτι πολύ σημαντικό. Άνοιξε δηλαδή ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των χωρών, όχι μόνο διμερός, αλλά νομίζω ότι ήταν και ένα μήνυμα προς ολόκληρη την περιοχή. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν πιστεύουμε ειλικρινά πως η διαδικασία διεύρυνσης είναι κάτι που πρέπει να δούμε και από την γεωπολιτική οπτική γωνία, καθορίζοντας και εκεί κριτήρια. Η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με την επιτάχυνση της διαδικασίας προκειμένου τα Δυτικά Βαλκάνια κάνει να μπορέσουν να γίνουν μια περιφέρεια και πολιτικά και οικονομικά και από πλευράς ασφάλειας. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερη πνοή στην επιθυμία και τους στόχους αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτά που μόλις τώρα μας είπε ο Υπουργός Εξωτερικών σε μεγάλο βαθμό τα επιβεβαιώνω. Δηλαδή η Αλβανία πράγματι καταβάλει προσπάθειες και ήδη διαφαίνονται κάποια αποτελέσματα. Εμείς στηρίζουμε την Αλβανία εκ βάθους καρδίας. Εκεί όμως που εξακολουθούμε να βλέπουμε προβλήματα είναι στη συνεργασία ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα στο Κοινοβουλίο, δηλαδή στο επίπεδο ε, του πολιτικού πολιτισμού, στις σχέσεις μεταξύ κυβερνητικού κόμματος και αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να βρουν κάποιο καλύτερο τρόπο συνεργασίας και θα πρέπει με καλύτερο τρόπο ο καθένας να ασκεί τα καθήκοντά του. Και από αυτού υπάρχουν ε, πολλές ε, δυνατότητες για να συζητήσουμε. Όσον αφορά στο ταξίδι του ε, Πρωθυπουργού προς τη Σερβία, του κυρίου Ράμα, ε, αυτό το βρίσκουμε θετικό το ταξίδι και για τις δύο πλευρές. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης καταδεικνύουν ότι τόσο η κυβέρνηση της ε, Σερβίας όσο και η κυβέρνηση της Αλβανίας έχουν συμφέρον μιας αγαστής συνεργασίας και Επίσης έχουν ε, συμφέρον να υπάρχει και ανταλλαγή νέων ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί και τη βάση μιας ε, καλής ε, σχέσης στο μέλλον. Έτσι για να αναφέρω ενδεικτικά ένα παράδειγμα. Βλέπουμε ότι, όπως σας είπα, οι εξελίξεις ε, στην Αλβανία είναι θετικές, όπως ακριβώς αναφέρεται και στην έκθεση Επιτροπής. Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν ακόμα θέματα όπου υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά στον τομέα παραδείγματος χάρη της δικαιοσύνης, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης πιο συγκεκριμένα, στον τομέα του αγώνα κατά της διαφθοράς, στον τομέα της διαφανούς ε, διοίκησης. Εμείς θα στηρίξουμε προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς όσο καλύτερα μπορούμε θα στηρίξουμε όμως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θέλουμε να ελπίζουμε ότι το συντομότερο δυνατόν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, λέει ο κύριο ε, Ζλάτκο Λαγκούμτζια. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο-τρία βασικά θέματα που είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα που ονομάζεται Βοσνία και Αρσεγοβίνη. Καταρχήν, πώς έχουν τα πράγματα. Είχαμε σχετικά πρόσφατα την ε, έκθεση πρόοδου και πριν από δύο μήνες ε, είχαμε εκλογές. Ελπίζουμε ότι θα θα σχηματιστεί η κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την προηγούμενη φορά. Σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε τη ε, βοσνιακή κυβέρνηση, όταν αναλάβει τα καθήκοντά τη, ε, θα ήθελα να πω ότι όλες οι πλευρές προσπαθούν να δημιουργήσουν ε, συμμαχίες και συνασπισμούς σε όλα τα επίπεδα, οντοτήτων, περιφερειών και σε κρατικό επίπεδο. Και είχαμε την πρωτοβουλία Βερολίνου, Λονδίνου, Βρυξελών μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε την Άνοιξη με πολλές εκδηλώσεις ε, και τα σημαντικά αποτελέσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών τον Απρίλιο στο Λουξεμβούργο. Τότε η Βοσνία και Ερζεγοβίνη πήρε προτάσεις ε, για το τι θα έπρεπε να κάνει στην περίοδο αυτή και μετά τις εκλογές. Τώρα, η πρωτοβουλία που έχουμε επιτάπητος ε, είναι ευπρόσδεκτη από όλου και δίνει τρει νέε προτεραιότητε στη νέα κυβέρνηση. Ευελπιστούμε ότι η νέα κυβέρνηση θα σχηματιστεί το συντομότερο δυνατό και δεν είναι το θέμα ποιο θα λάβει μέρο στην κυβέρνηση, αλλά ποια θα είναι η οικονομική και κοινωνική πλατφόρμα και πολιτική πλατφόρμα αυτή τη νέα κυβέρνηση. Ελπίζουμε τρει να είναι οι βασικέ προτεραιότητε τη νέα κυβέρνηση. Το κράτο δικαίου, δηλαδή εστίαση στο, στο διαρθρωμένο διάλογο και στις μεταρρυθμίσεις ε, της δικαστικής εξουσίας, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, δεύτερη προτεραιότητα οικονομική διακυβέρνηση και σύμφωνο για την ανάπτυξη και μάλιστα είχαμε εκτενείς διαβουλεύσεις ε, με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, μη κυβερνητικέ οργανώσει, επιχειρηματικού κύκλου, κοινωνία των πολιτών και εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτο πυλώνας τη νέα μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η μεταρρύθμιση τη δημόσια διοίκηση. Μάλιστα στον ανακοινωθέν του Υποσυμβουλίου Εξωτερικών του Απριλίου αναφέρεται και το θέμα αυτό. Μία ε, δημόσια διοίκηση θα αποτελέσει τη βάση για ένα εύρυθμο κράτος και η υπόθεση Σέιδιτς Φίντζη επίσης πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό, αλλά να μην μπλοκάρει τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και, και το κράτος δικαίου. Άλλο σημαντικό θέμα και η προτεραιότητα είναι η περιφερειακή συνεργασία. Κατά τη γνώμη μας, η περιφερειακή συνεργασία ε, των 6-7 χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ε, είναι σήμερα ακμεότερη από ποτέ καλύτερη από ότι τα τελευταία 5, 10, 20 χρόνια όσο και να ανατρέξετε. Και μάλιστα σημαντική όθηση ε, δόθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη Συμφωνία της Θεσσαλονίκης επί ελληνικής προεδρίας. Τότε είχαμε συνεδρίαση και με τους Υπουργούς Εξωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων και χάραξη της νέας ε, διαδικασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και στο πλαίσιο αυτό η περιφερειακή συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Η περιφερειακή συνεργασία προωθήθηκε και με τη διαδικασία του Βερολίνου ή τη συνεδρίαση του Βερολίνου με συμμετοχή πρωθυπουργών, υπουργών οικονομικών και υπουργών εξωτερικών και αυτή η συμφωνία θα πρέπει να ενισχυθεί στο μέλλον. Εμείς ε, έχουμε συναντηθεί τόσο συχνά τα, τον τελευταίο καιρό που θα έλεγα ότι οι παρακαθήμενοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους έρχομαι πιο συχνά σε επαφές το τελευταίο καιρό. Θα έλεγα ότι περισσότερο βλέπω εκείνους παρά τον εαυτό μου. Επίσης, ε, περιμένουμε με ανυπομονησία την επικείμενη επίσκεψη στο Σαράγεβο της Αντιπροέδρου Μογκερίνη και του Επιτρόπου Χάν. Και Είναι σημαντική αυτή η επαφή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι και καλή ευκαιρία για τους ε, ηγέτες της Βοσνίας Αρζεγοβίνης να καθίσουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και να μην πάει χαμένη η νέα πρωτοβουλία Βερολίνου, Λονδίνου ή Βρυξελών ή ευρωπαικη Ένωσης ή ε, να μην χαθεί αυτή η πρωτοβουλία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα να έχουμε σήμερα τη συζήτηση αυτή με τους Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων των Δυτικών Βαλκανίων. Πρόκειται για μια κοινή πρόκληση που έχουν μπροστά τους για να προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι εισηγητής για τη Βοσνία, οπότε οι ερωτήσεις μου απευθύνονται κυρίως στον κύριο Λακούμτσα. Η πρώτη έχει να κάνει με την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά τις εκλογές της Δευτέρας Οκτωβρίου που μας πέρασε. Θέλω να ξέρω λοιπόν πού βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας κυβέρνησης. Ελπίζουμε οι αρχές να εγκαθιδρυθούν ε, πολύ γρήγορα στη χώρα ο Πρωθυπουργό είπε ότι ελπίζει πως η διαδικασία διαπραγματεύσεων θα κρατήσει λιγότερο από ό,τι την προηγούμενη φορά, αλλά θέλω να ξέρω, πέρα από αυτά τα οποία παρακολουθούμε στον τύπο για τις συζητήσεις που γίνονται, στην πραγματικότητα πού βρίσκεται η διαδικασία προκειμένου να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Θέλω επίσης να γνωρίζω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα συνένεσης, να προκύψει συνένεση δηλαδή, για την ε, ημερήσια διάταξη και την ατζέντα όσον αφορά την ε, διαδικασία ένταξης της χώρας. Τα τελευταία που είπε ο Πρωθυπουργό όσον αφορά την γερμανοβρετανική πρωτοβουλία. Μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να καταλήξουν σε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Κατάλαβα ότι υπήρχε μια φυσιμία ε, στα λόγια του Πρωθυπουργού προς το τέλος. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά πιστεύω ότι οι χώρες πρέπει να συντονιστούν για να προχωρήσουν τόσο σημαντικές πρωτοβουλίες. Και γι' αυτό εύχομαι και εγώ ευρωπαϊκή συνένεση σε όλες τις χώρες μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πιστεύω εγώ ότι μπορούμε για πολύ καιρό ακόμα να παραμένουμε μέσα σε αυτήν την αμφισημία σε σχέση με τη νέα πρωτοβουλία. Αν πετύχαινε αυτό θα ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την δέσμευση της χώρας στον ευρωπαϊκό δρόμο, γιατί προς το παρόν η χώρα δεν, έχει, δεν είναι πια δεσμευμένη, είναι σαφές αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόκ και ευχαριστώ κύριο Σποπόσκη για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να συζητήσουμε με τους συναδέρφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφερθώ στο πλαίσιο. Αναφερθήκατε στη Θεσσαλονίκη και πιστεύω και εγώ την μεγάλη ενθάρρυνση για όλους μας το ότι δεν έχει ξεχαστεί δηλαδή η διαδικασία και ότι εξακολουθούμε να προχωράμε με τις ίδιες αρχές. Υπάρχει βέβαια και ένα εθνικό πλαίσιο. Η Μακεδονία, λέει ο μιλητής, είναι μια χώρα η οποία έχει υπογράψει συμφωνία στα θεροποίησης εδώ και λίγα χρόνια. Ήδη από το 2005 είχαμε την πρώτη σύσταση για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις το 2009. Είμαστε έξι χρόνια μετά και το μπαλάκι βρίσκεται στις χώρες μέλη και στην Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά τα μηνύματα είναι θετικά και πιστεύω ότι θα έπρεπε να τα δούμε στο πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα λυθεί απόφαση για νέα προσχώρηση. Ε, δεν νομίζω ότι είναι τραγικό γιατί αντικατοπτρίζει στο κάτω-κάτω την πραγματικότητα στις χώρες μέλη. Και δεν θα έπρεπε να το δούμε σαν κάτι τραγικό, από πλευράς των ε, Δυτικών Βαλκανίων, γιατί και αυτές οι χώρες πρέπει να προχωρήσουν οικονομικά και να προσαρμοστούν στο σύστημα στο οποίο θα αντιμετωπίζουν ε, προσχωρώντας. Δεύτερον, επικεντρωνόμαστε στον διάλογο υψηλού επίπεδου, έτσι όπως τον όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι κάτι που ισχύει για όλες τις χώρες, συνδυνάμει υποψήφιες χώρες της περιοχής τα κεφάλαια 23-24, τα οικονομικά, το κράτος δικαίου, τα μέσα ενημέρωσης, η διαφάνειά τους δηλαδή, η διαφήμιση, πολιτικό πλαίσιο, οι σχέσεις μεταξύ των διαφέρων φορέων και μετά υπάρχουν και οι εκλογικές συστάσεις από τον ΟΑΣΕ και από τον ΟΜΕΝΕΤΝ. Έχουμε ένα ειδικό κεφάλαιο το οποίο ονομάζεται «Σχέσεις καλής γειτονίας». Πρέπει βέβαια να το αποκωδικοποιήσουμε λιγάκι γιατί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχουμε καλές σχέσεις γιατί με όλες τις χώρες που δεν είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Τώρα για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δύο με την Βουλγαρία, έχουμε ένα καλό κανάλι επικοινωνίας και πιστεύω ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι θετικό, αλλά ο λόγος για τον οποίο υπάρχει το κεφάλαιο αυτό για τις καλές σχέσεις γειτονίας είναι η Ελλάδα. Και είναι το όνομα το οποίο ε, χρησιμοποιείται και υπάρχει μια επιπλέον, ένας επιπλέον όρος για να λυθεί αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτά τα πλαίσια δεν δείχνει ότι έχουμε κακές σχέσεις, γιατί οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Μακεδονία, λέει ο είναι πραγματικά εξαίρετες. Οικονομικά έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο των Σκοπίων από την Ελλάδα. Επίσης εμπορικό εταίρος σημαντικός είναι η Ελλάδα με εισαγωγές-εξαγωγές και έχουμε και πολλούς από τη χώρα μας που πηγαίνουν στην Ελλάδα για διακοπές. Καλέ σχέσει λοιπόν. Βέβαια το πολιτικό πλαίσιο είναι διαφορετικό και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια παραπάνω δέσμευση που λείπει προ το παρόν για να ξεπεραστεί και αυτή η πρόκληση, η δυσκολία. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με τα προηγούμενα, με το παρελθόν, το πλαίσιο και τις μεταρρυθμίσεις μας τώρα, είναι βέβαια οικονομικός παράγοντας. Έχουμε καλές επιδόσεις βάσει της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τριακοστή θέση, καλή θέση. Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ κοντά στα κριτήρια του Μάστριχτ, κάτι το οποίο δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Επίσης, όσον αφορά ε, το χρέος, είμαστε σε καλή κατάσταση. Χωρίς να θέλω να πω βέβαια ότι αυτό αντικατοπτρίζει την κατάσταση ολόκληρη την περιοχή, γιατί φυσικά η κάθε χώρα βρίσκεται στο μισό του ΑΕΠ, του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να καλύψουμε την απόσταση. Θέλω επίσης να πω ότι το πιο βασικό μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε σήμερα είναι να έχουμε περισσότερη αξιοπιστία στη διαδικασία και να προσδοκούμε αποτελέσματα από τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες. Γιατί τότε μπορούμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για προσχώρηση και να έχουμε στη συνέχεια μια περίοδο κατά την οποία να μπορούμε να προσαρμοστούμε στα όσα περιμένει από μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια να ληφθεί απόφαση για προσχώρηση. Ευχαριστώ και είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέω κύριος Βάγκλ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους καλεσμένους μας ότι οι φιλελεύθεροι είναι αναφανδόν υπέρ της διαδικασίας διεύρυνσης και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες που εκπροσωπείται. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, επιτρέπουμε να επικρατήσουν οι φόβοι που μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία διεύρυνσης. Και δεν θα ανάψει κόκκινο φως ε, στη διαδικασία διεύρυνσης. Ε, πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτή να σταματήσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών μας ενέφερε τις επιτυχημένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γιατί μειώνεται η ανεργία στη χώρα και το χρέος, το δημόσιο χρέος είναι σχετικά χαμηλό. Πολύ ωραία όλα αυτά. Η Μακεδονία είναι στη σωστή άγουσα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια προβλήματα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική στη διαθέτηση των εκκρεμωτήτων της. Είναι απαράδεκτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έκτη συνεχή χρονιά να συστήνει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και ακόμη να μην έχει πραγματοποιηθεί αυτή η έναρξη. Ακριβώς επειδή εκρεμεί το ζήτημα του ονόματος της χώρας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να επιδιώξουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη διαθέτηση αυτού του ζητήματος και ευελπιστώ ότι η νέα εκπρόσωπος ε, θα είναι πιο φιλόδοξη στο θέμα αυτό και πιο αποτελεσματική. Θεωρώ ότι οφείλουμε να ρυθμίσουμε το συντομότερο δυνατό αυτή την εκκρεμότητα και να, μάλιστα να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, και πριν την λύση του ζητήματος του ονόματος. Πιστεύω ότι παρόλα αυτά και παρά το, το ζήτημα του ονόματος η Μακεδονία θα πρέπει να ξεκινήσει τις ανταξιακές διαπραγματεύσεις. Φυσικά θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης και ελευθεροτυπίας και να εφαρμοστεί η Συμφωνία της Οχρίδας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην Βουλή. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να υπομιστούν τις ευθύνες τους για το μέλλον της χώρας. Και η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα, αλλά και η αντιπολίτευση θα πρέπει να αναλάβουν το τμήμα των ευθυνών που τους αναλογεί. Γιατί έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα πρέπει να λειτουργεί και η Μακεδονία. Γιατί εξαιτία αυτή τη αναποτελεσματικότητα ε, η Μακεδονία βρίσκεται σε πολιτική κρίση αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Ελμαρ Μπρόκ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που καλέσετε μένα και άλλους φίλους από την περιοχή για να ανταλλάξουμε απόψεις ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια και για τη διαδικασία διεύρυνσης. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω τα εξής σύντομα. Καταρχήν, θα ήθελα να ξεκινήσω επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες αλλαγής των σχέσεων ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς της περιοχής. Αυτή η αλλαγή των σχέσεων είναι και μετρήσιμη και ορατή. Ε, το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ ε, καθήμενη μπροστά σας ε, αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για το ότι πράγματι έχουν αλλάξει σχέσεις από εχθρικές, έχουν μεταφραστεί σε φιλικές, από μια ασταθή περιοχή είμαστε πλέον σταθεροί, υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ε, κυβερνήσεις, τους λαούς και τις οικονομίες και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτά, αυτή η αλλαγή και αυτά τα δείγματα υπονοούν σταθερότητα, αλλά για να είμαστε ειλικρινεί, αυτές οι αλλαγές δεν θα είχαν λάβει χώρα αν δεν υπήρχε η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίζει την περιοχή μέσα από τη διαδικασία διεύρυνσης, ε, την παροχή ε, τεχνικής ε, και οικονομικής βοήθειας και, και άλλου είδους βοήθειας. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε στο να βελτιωθεί η περιφερειακή συνεργασία, να διευκρινθεί η επίλυση πολλών ε, εκκρεμουσών υποθέσεων. Και είμαστε ευγνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας στήριξαν επειδή είμαστε όμως και πολιτικοί και εκπροσωπούμε τους λαούς μας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Στην περιοχή μας επικρατεί άποψη ότι πέρα από άλλες προκλήσεις, η περιοχή πλέον βρίσκεται ε, σε ένα status quo, σε μια κατάσταση που δεν αλλάζει. Και αυτό είναι απειλή. Δεν λέω ότι δεν σημειώσαμε πρόοδο, σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο. Όμως ε, είναι πολύ σημαντικό το να συνεχίσουμε να χαίρουμε τις υποστήριξή σας. Το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με, την ευρωπαϊκή, με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμένει πολύ σημαντική για όλες τις χώρες και για την κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου. Τα τελευταία 7 χρόνια μετά την εξαρτησία είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε μια ισχυρή, ένα ισχυρό πολιτικό πολυεθνικό ε, κοσμοπέδιο. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Εγώ μιλώ ως πολιτικός, εκπροσωπώ το κόμμα μου και είμαστε υπεύθυνοι για να καταρτήσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο ε, θα περιλαμβάνει πέντε βασικές προτεραιότητες. Πρώτον, οικονομική διακυβέρνηση. Δεύτερον, κράτος δικαίου. Τρίτο, ευρωατλαντικό θεματολόγιο. Τέταρτον, ε, παιδεία, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της παιδείας, ε, καθοριστική σημασία σε αυτό. Και το πέμπτο είναι η υγεία, η κοινωνική ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το ότι το 2014 για το Κωσυφοπέδιο ήταν μια ιστορική χρονιά γιατί μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κωσυφοπέδιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψουμε συμφωνία σταθερότητας. Έχουμε ήδη μονογράψει αυτή τη συμφωνία και ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να υπογραφεί η συμφωνία και να αρχίσει η εφαρμογή της το συντομότερο δυνατόν.

Αυτό καταδεικνύει επικοδομητικές σχέσεις ανάμεσα στο Κοσμοπέδιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι θεωρήσεις, ελεύθερες θεωρήσεις. Αυτή τη στιγμή το Κοσμοπέδιο είναι μια απομονωμένη νησίδα. Οι πολίτες μας είναι μόνοι τους στην περιοχή. Ε, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε χωρίς ε, θεώρηση. Από τον Ιανουάριο έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις. Προφανώς και είναι μια τεχνική διαδικασία. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, όμως χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε την ισχυρή πολιτική βούληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας δοθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία και να μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες Σέγγεν χωρίς θεώρηση. Το τελευταίο θέμα που θέλω να αναφέρω έχει σχέση με την περιφερειακή πολιτική συνεργασία και τη συμφιλίωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία 4-5 χρόνια ήταν ο διάλογος ανάμεσα στο Κοσφοπέδιο και τη Σερβία. Το 2013 επιτύχαμε μία ιστορική συμφωνία και νομίζω τότε ο πρόεδρος Τάτσιτς και ο πρωθυπουργός Βούτσιτς διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο. Όμως επιτρέψτε μου εδώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής και να πω ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή μιας ιστορικής διαδικασίας, ε, που δεν είναι το τέλος. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να υπάρξει πλήρης ομαλοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, αυτό πόρο απέχει από την τελική κατάληξη. Ε, εμείς θεωρούμε ότι ο διάλογος μπορεί να ωφελήσει και τις δύο πλευρές, παράλληλα όμως πρέπει να υπάρχει και ένας ε, στρατηγικός συλλογισμός. το πού θα οδηγήσει ο διάλογος. Και εδώ θέλω να αναφέρω πέντε βασικά βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν στο διάλογο ανάμεσα στη Σερβία και το Κωνσταντοπέδιο κατά επόμενα έτη. Πρώτον, πλήρης εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μέχρι τώρα. Ε, θα πρέπει να μην υπάρξει απόκληση και αναθεώρηση αυτών στη διαδικασία εφαρμογής του. Δεύτερον, να αποσυναρμολογηθούν όλες οι κρατικές δομές της Σερβίας μέσα στο Κοσοπέδιο. Τρίτον, πλήρης ενσωμάτωση των Σέρβων του Κοσοπεδίου στο κράτος μας. Τέταρτον, πλήρη συμμετοχή του Κοσοπεδίου στο διεθνές σύστημα, δηλαδή να γίνουμε και μέλος των ΗΕ. Και πέμπτον, πρέπει να έχουμε αμοιβαία αναγνώριση. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η προσέγγιση ε, για το πώς μπορούν να προχωρήσουν οι σχέσεις με τη Σερβία προς την κατεύθυνση της πλήρους ομαλοποίησης. Με αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει το διάλογο, στόχος είναι δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες και για μας είναι πολύ σημαντικό να υπογραφεί ε, συμφωνία ειρήνης που θα περιλαμβάνει την αμοιβαία αναγνώριση, τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων και την δρομολόγηση διαδικασίας ε, συμφιλίωσης ανάμεσα στις κοινωνίες μας. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, έχουμε σαφές θεματολόγιο και νομίζω την επόμενη εβδομάδα που θα εγκατασταθεί η νέα κυβέρνηση θα ξεκινήσει και η επόμενη φάση του διαλόγου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ εκ μέρου τη πολιτική μου ομάδα. Εδώ δεξιά είμαι, αν κάποιο θέλει να στρέψει το βλέμμα του, ή μπορείτε να με δείτε και στην οθόνη να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας από τις έξι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα χθε και τον Επίτροπο Χάν και την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη να διευκρινίζουν ότι η διαδικασία διεύρυνση θα συνεχιστεί με την ε, φόρα και την ισχύ όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Και ε, ελπίζω η αρχική δήλωση του κ. Γιούγκερ να μην αποθαρρύνει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα τάσσονται αναφανδών υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας διεύρυνσης. Εγώ θα μιλήσω για το Κόσοβο, το Κωσυφοπαίδιο, γιατί είμαι εισηγήτρια για τη σχετική έκθεση. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που αισθάνθηκα το τελευταίο εξάμεινο. Δημιουργήθηκε μια πολιτική αποτελμάτωση εξαιτία τη αδυναμία σχηματισμού κυβέρνηση. Ε, χαίρομαι που θα κλεγούν την επόμενη εβδομάδα και ο Πρόεδρος της Βουλής ε, και θα ορκιστεί και η νέα κυβέρνηση. Θα δώσω και εγώ το παρόν και χαίρομαι ιδιαίτερο που ενώ αρχικά δεν, είχα, δεν το είχα προγραμματίσει θα γίνω και εγώ μάρτυρας αυτής της δημιουργίας πρόοδου στο Κωσυφοπαίδιο. Ε, οι τελευταίες εκλογές στο Κωσυφοπαίδιο ήταν πολύ καλές ε, και το αποτέλεσμα έδειξε ότι ο λαός ψήφισε για αλλαγή και ευελπιστώ ότι η νέα κυβέρνηση θα επιφέρει τις νέες αλλαγές που προσδοκεί ο λαός του Κωσυφοπαιδίου. Μιλήστε για πολύ σημαντικά θέματα, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Α μην ξεχνούμε ότι έρχεται ο χειμώνα και στο Κωσυφοπαίδιο και η κατάσταση τη ενέργεια ε, θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τη νέα κυβέρνηση θα πρέπει ε, να αυξήσετε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και να μην στηρίζετε αποκλειστικά και μόνο στον άνθρακα που είναι επιζήμιο για την υγεία και να μειώσετε και την ενεργειακή σα εξάρτηση. Ε, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, ε, κράτο δικαίου και η κατάσταση των μειονοτήτων. Μερικέ εθνοτικέ μειονότητε, αλλά η Ρωμά, η Αιγύπτιοι, Ασκάλοι, ε, Γοράνη και άλλε μειονότητε δεν χαίρουν των δικαιωμάτων του, δεν μπορούν να τα ασκήσουν πλήρω και υπάρχει βελτίωση, αλλά περισσότερη εφαρμογή των συμφωνιών και καλύτερη εξασφάλιση των μειονοτήτων. Τώρα, ως προς το διάλογο. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είναι παρόντες σήμερα εδώ και οι δύο Υπουργοί τη Σερβία και το Κωσυφοπεδίου και θεωρώ ότι η πρόοδο αυτή είναι πολύ σημαντική για την εξομάλυση της κατάστασης και την ενίσχυση τη περιφερειακή συνεργασίας. Ευελπιστώ ότι και η Σερβία και το Κωσυφοπέδιο θα εφαρμόσουν τις υποσχέσεις τους ε, και τη συμφωνία για το διάλογο. Ελπίζω πολύ σύντομα να μπορώ να τηλεφωνώ στο κοσυφοπέδιο με ένα ειδικό κωδικό ε, κοσυφοπεδίου και όχι μέσω κωδικού Σλοβενίας ή Μονακό. Νομίζω ότι αυτό θα είναι σύμβολο των αλλαγών που θα λάβουν χώρα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που βρίσκει σύμφωνα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πλήρης εξομάλυση των σχέσεων Σερβίας-Κωσυφοπεδίου. Και τέλος, πολύ εύστοχα αναφέρατε και το θέμα της κατάργησης των θεωρήσεων. Η Τάνια, η Τάνια Φαγιόν ήταν αρμόδια για το θέμα αυτό στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Είναι παρούσα και στη συνεδρίαση. Είναι πολύ σημαντική η κατάργηση των θεωρήσεων ώστε να μπορούν και οι κάτοικοι του Κωσυφοπεδίου και οι πολίτε του Κωσυφοπεδίου να μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην εξακολουθούν να είναι οι μόνοι υπήκοοι χώρε που δεν μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ναι, αλλά αν μακρηγορείτε θα πάρει πολύ χρόνο και για το κοσυφοπαίδιο να υλοποιήσει αυτό το στόχο. Igor Λουξίτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωβουλευτές όντως. Όλα αυτά που λέτε αποτελούν μαρτυρία για την ε, μεγάλη δέσμευση των χωρών σας στο δρόμο προς την Ευρώπη. Δείχνετε ότι θέλετε να μοιραστείτε όλες τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Εθνών. Η οικονομική διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου είναι πράγματα τα οποία όντω πρέπει να κάνετε στο επόμενο στάδιο. Προκειμένου να μπορέσετε να τηρήσετε τις υποχρεώσεις σας για να ενταχθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται και για την οικονομική ανάπτυξη, πρόκειται για την ασφάλεια κλπ. η επίσκεψη του Επιτρόπου Χάν στο Μαυροβούνι δείχνει σε εμά ότι υπάρχει δέσμευση και από τη δικιά σας την πλευρά και ότι όντως παρακολουθείτε τις πρόοδους που κάνουμε. Επιτρέψτε μου να επενθυμίσω ότι προς το παρόν έχουμε κλείσει δύο κεφάλαια και έχουμε να ανοίξει άλλα δέκα και δουλεύουμε δραστήρια προκειμένου να ανοίξουμε και άλλα κεφάλαια βάση των επιτευγμάτων μας. Αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις που μας περιμένουν, αλλά είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε μεταρρυθμίσεις με απτά αποτελέσματα στο κράτος δικαίου και την οικονομική διακυβέρνηση. Όσον αφορά το κράτος δικαίου, βρισκόμαστε στη διαδικασία προσαρμόζοντας τα προγράμματα δράσης μας στα κεφάλαια 23 και 24 και θέλουμε ενισχυμένο έλεγχο και αξιολόγηση των επιτευγμάτων μας όσον αφορά την χρηστή διακυβέρνηση. Οι αξιωματούχοι μας ευθυγραμμίζονται στις προδιαγραφές σιγά σιγά και όλοι οι θεσμοί και όλα τα όργανα φροντίζουν γι' αυτό. Φροντίζουμε επίση για τη λογοδοσία, για την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, για την καταπολέμηση τη διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνεται και θα εγκριθεί τις επόμενες εβδομάδες, αφού βεβαίως έχουμε συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή. Όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και εδώ βελτιώνουμε το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται τα μέσα ενημέρωσης, φροντίζοντας να υπάρχουν ηθικές προδιαγραφές. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν το 2014 λύνονται σιγά σιγά και ξέρουμε ποιες είναι οι νέες υποθέσεις που έχουν προκύψει. Συνεργαζόμαστε με τη γραμματεία του ΑΣΕ στην ε, Βιέννη και την προσωπία τους στο Μαυροβούνι όσον αφορά τη δημοσιογραφία και προσπαθούμε να τηρήσουμε τον κώδικα διοντολογίας και ηθικής για τους δημοσιογράφους. Βάσει τώρα του οικονομικού προγράμματος που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2014 για νέα μέσα, όπως είναι τα ετήσια προγράμματα μεταρρυθμίσεων, είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει στη χώρα και προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Περιμένουμε περισσότερη οικονομική στήριξη από την άλλη μεριά, από την Ευρώπη για την περιοχή, για να βελτιωθούν οι υποδομές. Γιατί έτσι μπορεί να υπάρχει καλύτερη σύνδεση στην περιφέρεια μεταξύ των χωρών μας και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Το συμφέρον μας είναι κοινό υπέρ της Ευρώπης. Δεν θέλουμε μόνο οικονομική ανάπτυξη, αλλά θέλουμε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και τη μεταναστευτική πίεση. Θέλουμε περισσότερες προσπάθειες από την περιοχή για να αντιληφθούμε καλύτερα τα θέματα σταθερότητας και συνεννόησης στην περιφέρεια. Εμείς προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, να βελτιώσουμε επίσης το ε, επιχειρηματικό πλαίσιο και περιβάλλον. Υπογραμμίζω ότι όσον αφορά την έναρξη τον Ιούνιο 2014 των διαπραγματεύσεων για την κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας, προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε τις πολιτικές μας με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να αποφελθώ από την ευκαιρία αυτή επίσης για να σημειώσω εδώ την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποτελεί έναν πολύ βασικό εταίρο για μας στην διαδικασία ένταξής μας μας έχει βοηθήσει πολύ ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές με την κοινωνία των πολιτών, ακαδημαϊκούς και μας βοηθάει για την συμμετοχή όλων στην πορεία αυτή της διαδικασίας προς την ένταξη. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Μαυροβονίου τώρα για ένα λεπτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Αλμαρ με ευνηδία σα, Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Μαυροβουνίου σε αυτή την κοινή συνεδρίαση θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου για την παρουσία μου εδώ, να πω ότι ε, έχουμε ηγετική θέση στην ε, και στάση στην και με διαδικασία και είμαστε υπόδειγμα ε, πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να γίνονται φυσικά οι έλεγχοι και από την κοινωνία των πολιτών, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση ε, το κοινοβούλιο μας δηλαδή είναι παράδειγμα προς μίμηση για την περιοχή γιατί χωρίς ισχυρό κοινοβούλιο δεν μπορούν να, να υλοποιηθούν οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ε, Ήμουν 25 χρόνια στη Βουλή, έχουν αλλάξει χώρες, έχουν αλλάξει συστήματα, έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Οπότε μπορώ να αξιολογήσω τις μεταρρυθμίσεις, τη βελτίωση και να εντοπίσω και τα κενά και τις αδυναμίες. Πάντως η βάση για τη μεταμόρφωση, για τη μεταρρύθμιση είναι η ισχύς του Κοινοβουλίου. Νομίζω από αυτή την άποψη είμαστε από τις σταθερότερες χώρες των Βαλκανίων. Επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κοινοβούλια έχουν την ικανότητα να προωθήσουν τις κοινωνίες μας με παραγωγικό τρόπο και βάση για κάτι τέτοιο είναι το κράτος δικαίου. Η δικαιοσύνη είναι η βάση του κράτους και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες και ιδιαίτερα για τις ε, ε, νεοπαγείς δημοκρατίες. Έτσι μόνο θα αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία των πολιτών, την εμπιστοσύνη, την των πολιτών προς την ε, δημοκρατία και θα εξασφαλίσουμε και μια βιωσιμότητα του κράτους. Θα πρέπει η νομοθε... τα... τα νομοσχέδιά μας ε, να είναι αποτελεσματικά και με συνεργασία των κοινοβουλίων να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φάρος της περιοχής. Ε, αλλιώς ε, είμαστε ε, κάθε χώρα καράβια μέσα σε καταιγίδα και χωρίς ένα φάρο που να μας προσανατολίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτός ο φάρος και η σημασία της είναι πολύ πιο, σημαντική, πολύ πιο μεγάλη από ό,τι φαντάζεστε. Και έτσι θα, μπορούμε, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και τις προσδοκίες των πολιτών για περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη ασφάλεια και συνεργασία με τις άλλες δυνάμεις της περιοχής. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω μεγάλη πείρα στην Προεδρία της Βουλής, ίσως και είμαι και πιο μακρόβιος πρόεδρος Βουλής ε, στην Ευρώπη, το Μαυροβούνιο έχει μια σημαντική θέση, νομίζω, στην διαδικασία ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η δική μου ομάδα, η Εβδομάδα των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ε, παραμένει προσιλωμένη στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια όταν οι χώρες θα είναι έτοιμες. Ε, μέχρι τώρα είχαμε μια ιστορία επιτυχίας και καλωσορίζουμε τη Σερβία και την Αλβανία ως υποψήφιες χώρες ε, το Μοντενέγκρο και το Μαυροβούνι θα ακολουθήσουν και Λυπάμαι που δεν άνοιξαν οι διαπραγματεύσει με τη Μακεδονία κατά έκτη αυτή τη χρονιά παρά ε, το ότι είχαν προηγηθεί συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το Μαυροβούνιο, αυτή είναι η μόνη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια μέχρι τώρα η οποία προσωρινά έχει ανοίξει κάποια ε, κεφάλαια. Πρόκειται για τα θέματα εσωτερικών υποθέσεων ε, και δικαιοσύνη και έκλεισαν κάποια κεφάλαια επιστήμη και εκπαιδεία προ τιμή του. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με το πολλωμένο πολιτικό κλίμα ιδιαίτερα απολωμένο, κυρίως στο Κοινοβουλίο και αυτό παρεμποδίζει μερικές φορές την κοινοβουλευτική δουλειά που είναι απαραίτητη για να αφομοιωθεί το κοινοτικό κεκτημένο. Επίσης υπάρχουν κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη και την παρενόχληση των δημοσιογράφων. Δυστυχώς ε, η οικονομία πρέπει να είναι σταθερή, η ανεργία όμως είναι αρκετά υψηλή και υπήρξαν κάποιες ε, διαδηλώσεις για την οικονομία κατά τους τελευταίους μήνες. Το Μαυροβούνι προς τιμήν του έχει ήδη αντιμετωπίσει θέμα θύματα ε, των αλλοδαπών τζιχαντιστών που έχουν προσχωρήσει στον ISIS. Ε, μικρός αριθμός αυτών στο Μαυροβούνιο, αλλά υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός ε, στις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, κάτι που κανένας υπουργό Εξωτερικών μέχρι τώρα δεν έφτιαξε. Επίσης χαίρομαι που το Μαυροβούνιο που κινούμε την Αλβανία έχει προσανατολιστεί και έχει ευθυγραμμιστεί με τη δική μας τη θέση. Έχει επίσης υιοθετήσει, έχουν θετήσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης, Επίσης χαίρομαι ε, που έχει γη, στο Μαυροβούνι το θέμα του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Επίσης το Μαυροβούνι ελπίζει να επιτύχει το πράσινο φως από το ΝΑΤΟ για να προσχωρήσει κατά τους επόμενους μήνες. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια ουσιαστική αναγνώριση της συνεισφοράς του Μαυροβουνίου προς την περιφερειακή συνεργασία και την οικουμενική ασφάλεια. Ανακεφαλαιώντα, καλή αυτή η ιστορία του Μαυροβουνίου τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε βλέπουμε ε, αυτό που επιβεβαιώνεται που πολύ συχνά αναφέρεται, ότι το μικρό είναι και θαυματουργό. Ο κύριος Ντάτσιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση της Σερβίας πήρε την, το καθεστώς υποψηφίου και η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτη πολιτική προτεραιότητα της Σερβίας. Και από αυτή την άποψη είχαμε φέτος ιστορική πρόοδο, γιατί ξεκίνησαν επίσημα οι διαπραγματεύσεις, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πραγματικά ιστορική πρόοδος για τη Σερβία, μεγάλο ορόσημο και χαίρομαι που το θέμα της διεύρυνσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών. Η ενταξιακή προοπτική σίγουρα βοήθησε την βελτίωση των σχέσεων με τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Χάρη σε αυτή την ενταξιακή προοπτική, οι εκκρεμότητες στην περιοχή και τα ανοιχτά θέματα λύνονται με διάλογο. Και μάλιστα η ευρωπαϊκή προοπτική συνέβαλε και στο διάλογο και στη βελτίωση του διαλόγου Βελιγραδίου και Πρίστινας. Και αυτό έδειξε ε, την ε, έμπνευση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλύτερη συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια. Γίνεται πηγή έμπνευσης για μας. Και ε, είναι πολύ σημαντική ε, το πόσο δημοφιλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να πω ότι είναι πιο δημοφιλή η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Δυτικά Βαλκάνια από ό,τι σε μερικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσω είναι και λογικό κάτι τέτοιο. Προσδοκώ ότι το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ε, ευρωπαϊκής ε, ένταξης θα αγγίξει και τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Φυσικά δεν απάδομαι από τα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώσουμε για να γίνουμε πλήρως Φυσικά, κάθε χώρα θα πρέπει να κριθεί περιπτωσιολογικά, εξατομικευμένα, χωρίς ε, εσπευσμένο και επιβεβλημένο έξωθεν ρυθμό. Η, Ευρωπα... η Σερβία θα τηρήσει τα κριτήρια και από αυτή την άποψη προτεραιότητα μας είναι η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση η επικοδομητική πολιτική περιφερειακή συνεργασίας και αυτό το αποδεικνύει και η πρόσφατη συνεδρίαση που είχαμε στο Βελιγράδι μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών ε, της περιοχής. Η περιφερειακή συνεργασία και η οικονομική σταθερότητα είναι το κοινό μέσο για την υλοποίηση το, του κοινοτικού κεκτημένου και την πλήρωση των κριτηρίων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ολοκληρώσει το 21ο κεφάλαιο, ε, έχουμε ανοίξει 10 κεφάλαια και ελπίζουμε ότι θα τα ολοκληρώσουμε το πρώτο εξάμεινο του επόμενου έτους. Ε, θα πρέπει να κρατήσουμε αμύωτη τη δυναμική ε, των ανταξιακών διαπραγματεύσεων και η πρόοδος δείχνει ότι έχουμε πραγματικά διοικητικές ικανότητες και ότι είμαστε έτοιμοι σχετικά σύντομα να εστερνιστούμε και να εφαρμόσουμε το κοινοτικό κεκτημένο. Επίσης, τα κράτη-μέλη περιμένουν από την Σερβία ε, εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για το κρατοστικαίο, τη δημόσια διοίκηση, την ελευθερωτυπία, και την επίλυση του δημοσιονομικού ελλείμματος ή την όθηση και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Εμείς σε αυτή την περίοδο θα προσπαθήσουμε να συγκλίνουμε την πολιτική μας ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το άρθρο 10 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Το, την 1η Ιανουαρίου η Σερβία θα αναλάβει πολύ σημαντική ευθύνη, την Προεδρία της ε, ΟΑΣΕ που είναι πολύ περίπλοκο και λεπτό θέμα της ε, δέσμευσής μας. Βασικό, ε, βασική πρόκληση να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί σε όλα τα θέματα της ΟΑΣΕ και κατά την συζήτηση του θέματος της Ουκρανίας που σίγουρα θα βρεθεί στο επίκεντρο της ημερής σας διάταξης θα πρέπει να φροντίσουμε να συμβάλλουμε στην ε, επίλυση της κρίσης και τις δραστηριότητες αυτές θα τις ε, συνεχίσουμε και κατά διάρκεια της Προεδρίας μας ε, στην ΟΑΣΕ. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η Ελβετία που ήταν η προκάτοχος στην Προεδρία και ελπίζουμε και η Γερμανία που θα προεδρεύσει τις επόμενες τρεις μέρες ε, στη Βασιλεία. Προτεραιότητες μας φυσικά είναι η ειρήνη, η εξομάλυση των σχέσεων και η ευημερία των λαών. Ξέρω ότι σκοπός τέτοια, τέτοιων συνεδριάσεων είναι ο καθένας να παρουσιάζει με το καλύτερο φως τον εαυτό του και να δίνει όσο πιο καλύτερη εντύπωση μπορεί. Από αυτήν την άποψη θα μπορούσα να μιλήσω για πολλή ώρα ακόμη. Αλλά έχουμε συνηθίσει ε, τέτοιου είδους ε, συνεδριάσεις και τέτοιου είδους ε, συναντήσεις. Εμείς σχεδόν συναντιόμαστε μεταξύ μας κάθε εβδομάδα. Έχουμε τακτικότητες επαφές. Θα πρέπει όμως να έχουμε επίγνωση και της πραγματικότητας, της κατάστασης επιτόπου και να μιλούμε ανοιχτά και σταράτα για τα θέματα αυτά. Είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε ειρήνη και σταθερότητα και είναι πολύ εύκολο να καταστρέψουμε κάτι που πολύ με μεγάλο κόπο χτίσαμε. Γι' αυτό όλοι όσοι συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες και εμείς από τα Δυτικά Βαλκάνια και εσείς ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν μιλάτε για την χώρα και για, τα δυτικά, για τις χώρες μας και για τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να ξέρετε γιατί μιλάτε. Προ, τις προάλλες μιλήσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Σέσελ, ε, για τη Σερβία. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να μιλάει για ό,τι θέλει αλλά η Σερβία δεν έλαβε μέρος, ούτε επηρέασε την απελευθέρωση του, του Σέσελ. Το δικαστήριο της Χάγης δεν ενημέρωσε καν την Σερβία για την απόφαση αποφυλάκησης του Σέσελ, όπως έγινε και με τους προηγούμενους κατηγορούμενους. Και μάλιστα 11 χρόνια κράτησε ε, η δίκη αυτή. Κράτησε πολύ περισσότερο από ότι η δίκη να ζει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μάλιστα δεν εξέφρασε κανείς παράπονα όταν ήταν ο Σέσελ στη Χάγη για την, για την απόφαση αποφυλάκησης και άρχισαν να διαμαρτύρονται τώρα που βρίσκεται στο Βελιγράδι ο Βόιτσλαφ Σέσελ. Εγώ προσωπικά δήλωσα πολλές φορές ότι ο Σέσελ ανήκει στο παρελθόν, ότι η Σερβία δεν υποστηρίζει την πολιτική του. Και δεν καταλαβαίνω τα σχόλια ότι η σερβική κυβέρνηση δεν έκανε κανένα σχόλιο για τον Σέσελ. Επίσης, θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν δικαιούται κανείς να κατηγορεί ή να διώκει τον Σέσελ για οτιδήποτε άλλο από ό,τι κατηγορείται και διώκεται στο δικαστήριο της Χάγης. Ούτε να κατηγορείται Σερβία. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλήθηκε με πολύ απογοητευτικό τρόπο στη σερβική κοινή γνώμη και δόθηκε πολύ αρνητική εντύπωση. Η Σερβία έχει αλλάξει. Η Σερβία δεν είναι ίδια σήμερα με την, το με την στιγμή που βγήκε ο Σέσελ από τη Χάγη. Πριν από μερικά χρόνια δεν θα ήταν εύκολο να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Σίγουρα πριν το 2011 δεν θα μπορούσαμε να καθόμαστε δίπλα-δίπλα ο Χότζα και εγώ. Και έχουμε συζητήσει πολύ μεταξύ μας πριν καταλήξουμε στην Συμφωνία των Βρυξελών θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι όλα αυτά δεν τα κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κάνουμε για μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτός σκοπός, είναι μέσο, γιατί αστερνιζόμαστε τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Όλα τα έκρεμη προβλήματα θα πρέπει να τα λύσουμε διμερώς. Γιατί δεν μπορούν η Σερβία και η Κροατία διμερώς να τα συζητήσουν. Και μάλιστα ε, λυπούμε που με αίτηση της Κροατίας ακυρώθηκε το ταξίδι του Κροάτη Πρωθυπουργού στο Βελιγράδι μετά την, το ψήφισμα για το ΣΕΣΕ. Και μπορείτε στην εφημερίδα Βέτσερνη Λίστη να διαβάσετε τις δηλώσεις που είχα κάνει για το ΣΕΣΕΛ. Πιστεύω λοιπόν ότι η Σερβία έκανε τεράστιες προσπάθειες ε, και έφερε και αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε συνεχώς να επιστρέφουμε σε μια σχέση προς τη, στη Σερβία που είχε νόημα πριν από 20 χρόνια. Αλλά σήμερα με την σημερινή κατάσταση δεν έχει νόημα αυτή η σχέση πια. Η κατάσταση έχει αλλάξει, η Σερβία έχει αλλάξει. Γιατί σήμερα που μιλήσατε για το κοσυφοπέδιο κανένας δεν μίλησε για την ανάγκη ε, σχηματισμού δικαστηρίου ε, και την ε, εκδίκαση εγκλημάτων πολέμου. Γιατί δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Γιατί και αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες μας. Εγώ δεν είπα γιατί απελευθέρωσε το δικαστήριο της Χάγης κάποιους Αλβανούς, Κροάτες, στρατιωτικούς διοικητές, ούτε μίλησα για την εκστρατεία κατά του κυριλικού αλφαβήτου που λαμβάνει η χώρα στην Κροατία. Όλα αυτά τα θέματα μπορούμε να τα λύσουμε διμερώς. Εγώ συμφωνώ ότι η πολιτική του Σέσελια θα πρέπει να στυλιτευτεί και να καταδικαστεί. Αλλά να μην καταδικαστεί η Σερβία, γιατί η Σερβία καταδίκασε αυτή την πολιτική. Και ακριβώς η πολιτική που επικράτησε στη Σερβία είναι πολιτική αντίθετη με αυτή του Σέσελ. Μίλησα περισσότερο, αλλά ακριβώ επειδή και εσεί ε, μιλήσατε εκτενώ για μα και μάλιστα ερήμην μα και την απουσία μα, ε, πήρα και εγώ το θάρρο να μιλήσω λίγο παραπάνω για τη Σερβία. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Ο κύριος Αλής ε, που είναι επικεφαλής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας είναι σήμερα στην Ουάσιγκτον και δεν μπορεί να λάβει το λόγο ως εισηγητής. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα πω ότι σε γενικές ε, γραμμές της εξελίξης της Σερβία τις κρίνουμε θετικές και πρόκειται για σταδιακή εφαρμογή των υποχρεώσεών της που απορρέει από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ασφάλειας. Αυτό λοιπόν είναι θετικό και όταν επισκέφτηκα τη Σερβία αποκόμισα την εντύπωση ότι υπάρχει σοβαρή βούληση να εφαρμοστούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, να δημιουργηθούν κάποιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης. Όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να προσαρμοστεί ένα σύστημα είτε πρόκειται για τον ε, νομικό, ε, δικαστικό τομέα, τη δημόσια διοίκηση, το συνταξιοδοτικό με όλα αυτά που συνεπάγεται σε δημόσια συζήτηση. Όμως έχω την εντύπωση σε συζητήσεις ε, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών ότι πράγματι υπάρχει η κατηγορηματική βούληση να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διαφθορά. Και επίση, είμαι σίγουρος ότι η Σερβία με επικοδομητικό τρόπο θα δεχθεί την ε, πρόσκληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεργαστεί στον μηχανισμό προστασίας πολιτών. Κυρίες και κύριοι, τα βήματα που έχουν γίνει στη Σερβία και στο Κοσφοπέδιο ελπίζω να, ελπίζω να συνεχιστούν. Συζήτησα και με τις δύο πλευρές και αποκόμισα την εντύπωση ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν σταδιακά να δρομολογήσουν εξελίξεις έτσι ώστε με την πάροδο των ετών να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα, κανένα πρόβλημα που να παρεμποδίζει τη διαδικασία διεύρυνσης. Και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να το στηρίξουμε αυτό. Πιστεύω ότι η Σερβία με τις παραδοσιακά καλές σχέσεις της με τη Ρωσία έχει πολλές δυνατότητες μέσω μιας ειρηνικής λύσης και το 2015 επειδή θα προεδρεύσει στον ΟΣΑ θα έχει ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Αυτό πρέπει να το στηρίξουμε. Γνωρίζουμε ότι στη Σερβία υπάρχουν πολλά εκκρεμή θέματα. Έθιξα το θέμα των μεταρρυθμίσεων, της διαφθοράς. Αλλά σας το είπα ήδη ότι εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι αποφασισμένοι να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Και εκεί στη Σερβία όπως και αλλού υπάρχουν πολύ σκληρές συζητήσεις όσον αφορά την κάθαρση από το παρελθόν και την αντιμετώπιση του μέλλοντος. Ο πρώτος καγκελάριος Γερμανίας, ο Κόνατ Αντενάου, είχε πει το εξή Η ιστορία υπάρχει για να εξάγουμε συμπεράσματα από την ιστορία και να βελτιώσουμε το μέλλον. Η ιστορία δεν πρέπει να υπάρχει απλά και μόνο ως μοντέλο και πρότυπο για το τι πρέπει να επαναλάβουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου εμείς οι πολιτικοί έτσι ώστε να δίνουμε θετική νότα στις διεργασίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμεθα λοιπόν στην κανονική μας συζήτηση και ως πρώτος θα λάβει το λόγο ο κύριος Πλένκοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί Υπουργοί. Εγώ στηρίζω τις φιλοδοξίες όλων των χωρών που παρίστανται στο να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου. Και θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν μπορούσαμε επιτέλους να ανοίξουμε τις ε, συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις ε, ένταξης της Μακεδονίας. Επίσης, ε, να σας πω ότι παρακολουθούμε το τι συμβαίνει στο Κοινοβουλίο της Μακεδονία. Μακεδονία και τη Αλβανία, αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βοσνία και η Σεγοβίνη βρίσκονται στην καρδιά των προτεραιοτήτων μα ε, κυρίω μετά τι εκλογέ τη 12 η Οκτωβρίου. Προσβλέπουμε στη δημιουργία τη ε, νέα κυβέρνηση, ε, όπου θα εκπροσωπούνται νόμιμα οι συντακτικέ οντότητε των χωρών αυτών. Όσον αφορά τώρα στα τελευταία σχόλια που αφορούν στα σχόλια του Ντάτιτς ε, που αναφέρθηκε στο ψήφισμα των, Ευρωμένων, ε, των, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ε, καταδίκες εγκληματιών. Θέλω να πω το εξή. Εχθές είδαμε τον Μπράμερτς, τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ζήτησε να ανακληθεί αυτή η απόφαση και το θέμα να ξανασυντηθεί στην Χάγη, στο δικαστήριο Κύριε Υπουργέ, μας είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Σερβία. Ελπίζω στη Σερβία να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και ευρωπαϊκές αξίες. Ο Σέσελ, σχετικά με την επιστροφή του, προέβη σε απαράδεκτες δηλώσεις και άρα ήταν απαραίτητο να υπάρξει απερίφραστη καταδίκη από τις αρχές της Σερβίας. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλετε να είσαστε αξιόπιστοι υποψήφοι, γιατί η διαδικασία ένταξη έχει σχέση και με την αξιοπιστία και αν θέλετε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δεν μπορείτε να γνωείτε ή να παραλείπετε, να καταδικάζετε μεγαλοστομίες που έχουν σχέση έστω και με πριν από 20 χρόνια. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετείτε με απόλυτη σαφήνεια επ' αυτού. εκτός μικροφώνου. Δυστυχώς γίνονται σχόλια εκτός μικροφώνου. Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στη δήλωση της Θεσσαλονίκης που στηρίζουμε πλήρως. Στις 28 Νοεμβρίου, λοιπόν, η Γαλλία μέσω του Υπουργού της Εξωτερικών Υποθέσεων υπενθύμησε ότι θεωρεί κυρίως την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προτεραιότητα για την σταθερότητα στην περιοχή. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιμένει πέντε χρόνια για τεχνικούς λόγους, είπατε. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε με ελπίδα και αποφασιστικότητα να εξετάζουμε την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη. Στο χρονικό αυτό διάστημα θέλουμε να προχωρήσουμε σε παραδειγματικού τύπου διαπραγματεύσεις. Εννοείται ότι χρειάζονται μακρές διαπραγματεύσεις και για την οργάνωση των διαπραγματεύσεων αυτών θέλουμε να καθορίσουμε προτεραιότητες. Έχουμε πάρει τα μαθήματα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά το παρελθόν. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς επαλήθευσης και συνεργασίας και μετά την ένταξη, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι ικανοποιητικό. Γι' αυτό και θέλουμε να αποφύγουμε την ένταξη χωρών που βρίσκονται πολύ μακριά ακόμα από τις καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να προσχωρήσουν χώρες που είναι έτοιμες να δεχτούν τους κοινούς κανόνες και να αποφεληθούν από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Για το σκοπό αυτό θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν αποτελεσματική δίκηση και ικανοποιητική δικαιοσύνη. Έχουμε τη συνήθεια να ανοίγουμε ε, διαπραγματεύσει από το κεφάλαιο για το κράτο δικαίου και την ε, λειτουργία τη δικαιοσύνη. Είναι θετικό αυτό. Σω θα μπορούσαμε να πάμε πιο μακριά και να προβλέψουμε ένα άλλο κεφάλαιο πριν ε, αρχίσουν οι συζητήσεις για αυτά τα δύο κεφάλαια ή πριν έχουν προχωρήσει αρκετά ώστε να ε, κλείνουν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα θέλαμε προτεραιότητες βασικινής λογικής, αλλά κυρίως να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική και θετική και δίκαιη ολοκλήρωση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω και εγώ να καλωσορίσω τους φιλοξενούμενους μας και να πω ότι σας στηρίζω στην διαδικασία σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω την πολιτική σας βούληση. Θα ήθελα όμως να κάνω τρία σχόλια, επιτρέψτε μου. Τρία σχόλια για όλες τις χώρες μαζί. Πρώτα απ' όλα υπάρχει διαφθορά. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αυτό όμως που είναι ακόμα πιο προβληματικό, πιστεύω, είναι το θέμα του πλουραλισμού και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Η πολιτική και οικονομική πίεση, οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους, ε, ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητες έρευνες για τέτοιου είδους θέματα. Πράγματα που δεν χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη κοινωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κάνετε κάτι παραπάνω για να έχετε ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πρέπει να δημιουργήσετε το σωστό περιβάλλον, γιατί οι δημοσιογράφοι κάτω από πίεση φυσικά δεν είναι κάτι καλό για δημοκρατικές λειτουργίες. Συναντήθηκα πρόσφατα με ακτιβιστές από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αγωνιστές για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ, για παράδειγμα. Η ομοφιλοφοβία πρέπει να ξέρετε ότι είναι κάτι σοβαρό και πρέπει και γι' αυτό να κάνετε κάτι. Υπάρχουν όλο και περισσότερες εκθέσεις για διακρίσεις που γίνονται, για επιθέσεις που γίνονται σε βάρος ατόμων ΛΟΑΤ και άλλων ευάλωτων ομάδων, όπως μέλη μειονοτήτων. Είναι πράγματα τα οποία βέβαια πρέπει να προσέχουν όλες οι χώρες, όχι μόνο εκείνες των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά του κόσμου ολόκληρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ελλάδα πάντα υποστήριζε ισχυρά την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως και η Προεδρία, έτσι και εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στην ευρωπαϊκή προπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και θέλουμε να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι κάτι απόλυτα συνδεδεμένο με τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιες χώρες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η διαδικασία και η συμφωνία του Ελσίνκη. Πρέπει να προσπαθήσουν μεταξύ άλλων για συμφιλίωση και για να αντιμετωπίσουν τις πηγές του αρνητικού εθνικισμού. Όσον αφορά το πακέτο διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζουμε το γεγονός ότι υπογραμμίζονται για παράδειγμα τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια και οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις όπως επίσης και οι καλές σχέσεις γειτονίες που αποτελούν προϋπόθεση για τη διαδικασία διεύρυνσης. Επίσης, στηρίζουμε την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσδιεύρυνση για τις χώρες προς ένταξη. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει όμως ε, μεικτά μηνύματα προς τα Σκόπια. Το θέμα του ονόματος δεν είναι άλοθη. Δεν πρέπει να είναι άλοθη για την έλλειψη μεταρρυθμίσεων από πλευρά της χώρας. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας αυτής, εφόσον τα ευρωπαϊκά κριτήρια καλύπτονται πλήρως, μεταξύ άλλων και οι πραγματικές καλές σχέσεις γειτενίε και το θέμα επίλυσης του ονόματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαι υπέρ τη πολιτική διεύρυνση, είμαι υπέρ των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ξέρω ότι είναι δυσχερή διαδικασία, για άλλε χώρε είναι πιο εύκολη, για άλλε πιο δύσκολη. Δεν θα ήθελα όμω κανένας να μείνει πίσω ή να εγκαταλείψει, γιατί η σταθεροποίηση και η σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων σημαίνει σταθερότητα για ολόκληρη την Ευρώπη. Παρατήρησα ότι ε, η αλαζονία, κύριε Ντάτσιτ δεν περνάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί μιλήσατε πολύ αλαζονικά και είπατε ότι εμείς ταυτίσαμε την Σερβία με τις δηλώσεις του Σέσελ. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Απλώς ζητήσαμε από την κυβέρνηση της Σερβίας να αποστασιοποιηθεί από τις δηλώσεις του Σέσελ. Γιατί γνωρίζουμε τι συνέβη στα Βαλκάνια, γνωρίζουμε την ιστορία. Μάλιστα ο κύριος Ντάτσιτς ήταν ε, από τη που δεν είναι, μήπως ήταν ε, στενός ε, συνεργάτης του Σέσελ θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από την πολιτική του Σέσελ Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, θέλουμε να αποκηρύξει η Σερβία την πολιτική του Σέσελ να, αποστασιοποιηθεί συγγνώμη από τις δηλώσεις του Σέσελ Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου και εμείς παρακολουθούμε τις προσπάθειες ε, των Δυτικών Βαλκανίων, όπως βέβαια και άλλοι συνάδελφοι. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους που βρίσκονται εδώ και να ευχαριστήσω και το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή που συνέταξαν αυτά τα πολύ χρήσιμα έγγραφα. Χρήσιμα για μας όταν συζητάμε για τη διεύνηση ε, με εκπροσώπους κοινή γνώμη να πω κάτι σχετικά με το έγγραφο εργασίας. Εδώ πρόκειται από μόνο του για πρόγραμμα και παραθέτω χώρες και ειδικέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές για σημαντικά θέματα που έχουν μέχρι τώρα μπλοκάρει την ε, πρόοδο. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά επόμενα 5-6 χρόνια. Αυτό να γίνει. Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, να ονοματιστούν όχι έτσι με ασάφεια αλλά με σαφήνεια και ε, να εξεταστούν και μετά να δούμε πώς ακριβώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει βοήθεια να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να μετρήσουμε επίσης και το πώς οι εν λόγω χώρες ε, θα προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν και αυτές τις προκλήσεις. Αυτά πρέπει να κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια αν δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο. Και ολοκληρώνοντας εύχομαι τα καλύτερα στις χώρες των Βαλκανίων, στην προσπάθειά τους για μετερθμίσεις και να μην ξεχάσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν για τη συμφιλίωση όχι μόνο ανάμεσα στις χώρες αλλά και μέσα στις χώρες ανάμεσα σε διαφορετικές εθνοτικές ομάδες και σε κάποιες χώρες επίσης συμφιλίωση στα κοινοβούλια ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ. εκ μέρους των εργατικών Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο λέει ο κύριο Κιρτσόκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί υπουργοί, σα καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω ρωτήσει προ τη Σερβία. Στα μέσα Οκτωβρίου, Σερβία-Ρωσία υπέγραψαν διάφορε συμφωνίε, ε, μνημόνια και πρωτόκολλα κατά την επίσκεψη του Πούτιν στο Βελιγράδι. Και μία συμφωνία αφορά στην τεχνική και στρατιωτική συνεργασία. Και μία άλλη συμφωνία για την αμοιβαία προστασία απόρριτων πληροφοριών. Η Σερβία υποσχέθηκε να μην εφαρμόσει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία και να προχωρήσει με τον αγωγό South Stream. Και έχουμε όμως ξεκινήσει εμείς διαπραγματεύσει με τη Σερβία. Μετά τις εκλογές ε, και τις, μάλλον, με μετά τις δηλώσεις του Πούτιν που έλαβαν χώρα εχθές, τι θα κάνετε, είστε πρόθυμοι να επιβάλλετε κυρώσεις στη Ρωσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να εκφράσω την στεναρή υποστήριξη της Σουηδίας προς τη διεύρυνση. Νομίζω γνωρίζετε όλοι σας ότι εμείς παραδοσιακά είμαστε υπέρμαχοι αυτής της ε, διεύρυνσης. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι ε, για τις υποψήφιες χώρες να σημειώσουν πρόοδο αυτό κυρίως αφορά χώρες ε, που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Για την περίπτωση τώρα τη δική μας, της Σουηδίας, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, να τίνουμε χείρα βοηθείας. Για μας υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να συνεργαστούμε με χώρες οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, να ακολουθήσουν ε, το δυτικό τρόπο ζωής και σκέψης. Σημαντικές λοιπόν αξίες να υπάρξουν, να τις στηρίξουμε. Παραδείγματος χάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η ισότητα, ο σεβασμός ε, των ΛΟΑΔ και μη διακριτική μεταχείριση. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να σας στηρίξουμε στη δουλειά σας όπως σας είπα, είμαστε στεναροί υποστηρικτές της διεύρυνσης και ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να καλωσορίσουμε περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν θα είσαστε έτοιμοι και όταν ε, θα έχουν καλυφθεί όλα τα απαραίτητα κριτήρια θα είσαστε ευπρόσδεκτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το στηρίζει ανεπιφύλακτα το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν λιγάκι κανείς ε, την έκθεση πρόοδου για τα Δυτικά Βαλκάνια, διαπιστώνει ότι για κάθε χώρα υπάρχει το κεφάλαιο 23 που επισημαίνεται που αφορά τον τρόπο διαβίωσης των ε, Ρωμά και των Ασκάλι. Γίνεται κάποια πρόοδος και αναφέρεται αυτή, αλλά σε μεγάλο βαθμό διαπιστώνουμε ότι οι Ρωμά ζουν σε άθλιες συνθήκες στις περιοχές αυτές. Δεν έχουν δικαίωμα σε παιδεία, ε, στέγαση, κοινωνικά συστήματα. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα έπρεπε ή θα παρακαλούσε τους υπουργού εξωτερικών να τοποθετηθούν σε αυτά τα θέματα, δηλαδή να μας πούνε τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες τους για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και επιτρέψτε μου και μία παρατήρηση προς τη γραμματεία της Επιτροπής μας. Είμαι ευγνώμων για τα έγγραφα που μας στείλατε για την προετοιμασία της Επιτροπής, όμως βλέποντας το έγγραφο εργασίας που γίνεται λόγος για τις προκλήσεις και τις δυνατότητες των Δυτικών Βαλκανίων, μόνο μία φορά αναφέρεται η περίπτωση των Ρωμά και μόνο για μία χώρα. Επιθυμούμε λοιπόν στο μέλλον το θέμα αυτό να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη επάρκεια. Η κυρία Μπέκ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά χαρά για μας να βλέπουμε εδώ να κάθονται κοντά έξι Υπουργοί Εξωτερικών μετά αυτή την αιματηρή διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Μια εποχή που τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά κοινός δρόμος προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, περικλεί και κινδύνους, διότι όπως ακούσαμε και χθες, η Ρωσία επιδιώκει την πρόθεση νέων γεωστρατηγικών συμφερόντων που έχουν ε, διατυπωθεί με μεγάλη σαφήνεια, κυρίως όταν έγινε λόγο για την παράταση ε, της ε, ομάδας U4. Μέχρι τώρα υπήρχε απόλυτη συμφωνία από αυτού και τώρα για πρώτη φορά ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι η Ρωσία τάσεται κατά της παρουσίας οποιασδήποτε διεθνούς δύναμης στη Βοσνία γιατί με τον τρόπο αυτό προωθείται η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Ερωτώ λοιπόν, μήπως ε, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για κάτι το οποίο ενδεχομένως τώρα δεν θέλουμε να δούμε. Και Έχω κατά νου τον κίνδυνο η Σπέρτσκα να διοργανώσει δημοψήφισμα και να θελήσει να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της όπως έγινε στην Υπετινιστερία, στην Απχαζία αλλά μην ξεχνάτε και στην Κρυμαία. Ε, κύριε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω ερώτηση προς τον αξιότιμο Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, αλλά επειδή δεν τον βλέπω εδώ, παρακαλώ να μου δοθεί αργότερα ο χρόνος ομιλίας. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ο πρόεδρος ομιλεί εκτός μικροφώνου και δεν ακούμε τι λέει. Λυπάμαι. Αντώνιος Ατσουμπάλης, παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Uh, Ευχαριστώ, Έλμαρ. Και συγχαρητήρια, συνάδελφοι. Θα ήθελα εκ μέρους της ε, Ουγγρικής Βουλής να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις ε, ομιλίες σας και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συνεδριάζουμε και γι' αυτό ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μπρόκ που οργάνωσε αυτή την συνεδρίαση με συμμετοχή των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Υπουργών Εξωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ μεστές και περιεκτικές οι παρεμβάσεις και μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές στο θέμα της διαθέτησης της κατάσταση των εθνοτήτων. Χαιρόμαστε και είμαστε πλέον προς τον κύριο Ντάτσης για τη διαδικασία επανασυμφιλίωσης ε, της ε, ουγγρικής ε, μειονότητας στη Σερβία. Και ευχαριστούμε θερμά και τους κυρίους Νίκολης και Ντάτσης, τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό. Ε, συμφωνώ με τις δηλώσεις του κυρίου Ντάτσιτς ε, και σίγουρα η περίπτωση Σέσελ χρήζει εξονυχιστικής ανάλυσης. Πώς το καλό επέστρεψε στην Σερβία χωρίς ε, απόφαση του δικαστηρίου. Επίσης για τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια μπορεί να επιδεινωθεί. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε η κυρία Μπέκ ότι η ρωσική η εξωτερική πολιτική προσπαθεί να αλλάξει τη στάση απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και φαίνεται ότι εντατικοποιείται η παρουσία της Ρωσίας ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και θα πρέπει ε, να προσέξουμε μήπως εμφανιστεί ριζοσπαστικό Ισλάμ μέσα στα Δυτικά Βαλκάνια. Τα κενά καλύπτονται. Υπάρχει αυτή η τάση να μην μένουν κενές περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην δημιουργηθούν κενά. Επίση, ο κύριο Γιούγκερ είχε πει ότι για μία πενταετία αποκλείεται διεύρυνση. Μου θύμισε την Άννα Σουχότσκα, την Πολωνέζα Υπουργό Εξωτερικών, που είπε ότι για μία δεκαετία ακούγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να περιμένετε πέντε χρόνια. Ελπίζω να μην είναι τέτοια τα πέντε χρόνια που θα περιμένει που θα περιμένει τα Δυτικά Βαλκάνια όπως περίμενε η Κεντρική Ευρώπη. Περιμένω από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το νέο κατεστημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρουν τρόπους για να κάνουν πιο θετικές δηλώσεις και πιο θετικές χειρονομίες προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Άλλωστε βρισκόμαστε στο κτίριο Γιώζεφ Άνταλ, πολύ κοντά στην 25η επέτειο των πρώτων δημοκρατικών εκλογών της Ουγγαρίας. Και θα ήθελα να θέσω και ένα ζήτημα. Φυσικά θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να ετοιμαστούν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για τη διεύρυνση, αλλά τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για τη διεύρυνση. Είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις αγκάλες μας και να προσκαλέσουμε αυτές τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι πρόβλημα ή μήπως είναι τμήμα της λύσης για την οικονομική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε και πνευματικά αλλά και οικονομικά και πολιτικά έτοιμοι να δεχτούμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω εκεί. Ε, θα έλεγα οι 7 υπέροχοι είναι το σωστός αριθμός. Πολύ χαίρομαι για αυτή τη διαδικασία διεύρυνσης. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αν δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, αμοιβαία κατανόηση και στήριξη. Αυτό πρέπει να υπάρχει και στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη της διαδικασίας. Πρέπει να καταλήξουμε σε λύσεις για τα προβλήματα που κρατούν καιρό και να ξαναδούμε την διαδικασία αυτή διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι πολύ πάντως για τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Το Μαυροβούνι, η Σερβία έχουν ανοίξει τις διαπραγματεύσεις, έχουν το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Αλλά υπάρχουν ε, προβλήματα που κρατούν, επιδεινώνονται κάποιες καταστάσεις στην Μακεδονία, λέει ο που δείχνουν τα πραγματικά προβλήματα. Στο μέλλον λοιπόν δεν πρέπει να τα δούμε αυτά σαν ένα διμερές πρόβλημα, αλλά σαν ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Βοσνία-Ερζεγοβίνη και εκεί έχουμε δει ότι η χώρα κάνει και πίσω βήματα σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις της στην πολιτική της. Πρέπει λοιπόν να ξαναμπεί στον ευρωπαϊκό δρόμο η χώρα με πρωτοβουλίες. Σερβία, πεδιο Σερβία, Αλβανία. Οι σχέσεις πρέπει ακόμα να βελτιωθούν. Είναι ζωτική σημασία για να διατηρηθεί ο δυναμισμός της ε, διαδικασίας. Στην ε, Μακεδονία, την Αλβανία υπήρξαν κάποια ποικοτάζ στην διαδικασία. Χρειάζεται και η ευθυγράμμιση επίσης των χωρών στις αρχές της κοινή εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εξηγηθούν καλύτερα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επόμενος ομιλητής. Δύο πράγματα. Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να ακούσω και να δω την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τα τελευταία χρόνια. Το τελευταία 25 χρόνια έχουν κάνει πραγματικά τεράστια πρόοδο. Βέβαια δυστυχώς ακούγονται και πράγματα που δεν είναι χρήσιμα. Ας το παραδεχτούμε. Πρέπει να λύσουμε πρώτα τα δικά μας τα προβλήματα, να μην ανακατευόμαστε με τον άλλον. Ο Σέσελ έχει την ιστορία κάθε χώρας μας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τα βάζουμε με το γείτονα Σέσελ, αλλά πρέπει να κοιτάμε πρώτα τις δικές μας περιπτώσεις. Το πώς βλέπει κανείς την ιστορία, τα ιστορικά γεγονότα, διαφέρει. Ιδιαίτερα οι γείτονες κοιτούν με διαφορετικό τρόπο τις καταστάσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πάντως, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε έναν λαό να δεχτεί την δικιά μας εκδοχή της ιστορίας, γιατί μετά από μερικές γενιές μπορούμε να έχουμε φτάσει και εμείς σε μια κατάσταση που να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Δεν μπορούμε πάντως σε 20 χρόνια μετά από όλη αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε να υποχρώσουμε κανένα γείτονα να δεχτεί τη δικιά μας εκδοχή της ιστορίας. Μετά από μερικά χρόνια μπορεί να γίνει, τώρα όμως δεν γίνεται. Πρέπει να ασχοληθούμε με τους εαυτούς μας, με το δικό μας κοινό μέλλον και όχι με το σκούρο παρελθόν μας. Ε, καταρχάς συμφωνούμε όλοι ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι ένας δρόμος ε, ο οποίος είναι χωρίς επιστροφή. Επιστροφή στα δεινά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες στην ε, πολύπαθη αυτή περιοχή. Τώρα ως ε, σκιώδης εισηγητής στο φάκελο του Μαυροβουνίου θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Μαυροβουνίου εάν έχουν επαρθεί κάποιες πρωτοβουλίες όσο αφορά το νομοθετικό πλαίσιο χρηματοδότηση των κομμάτων και όσον αφορά τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής εναντίον της διαφοράς. Και τέλος θέλω να υπογραμμίσω στον ε, Υπουργό Εξωτερικών της ε, ΦΥΡΟΜ ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση στο κλίμα των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών αλλά όσο αφορά την ονομασία, για να υπάρξει μια δίκαιη λύση, αυτή η λύση πρέπει να εδράζεται καταρχάς στην κοινή λογική και δεύτερο στην ιστορική πραγματικότητα των δύο αυτών χωρών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τους Υπουργούς Εξωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων που ήρθαν στη συνάντηση αυτή. Η Ρουμανία συνεχίζει να στηρίζει την ευρωπαϊκή προσχώρηση, την προσχώρηση δηλαδή όλων των χωρών που το επιθυμούν προκειμένου να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον τηρούν τα κριτήρια. Είναι και το κεντρικό στοιχείο το οποίο καθορίζει εξάλλου και το ρυθμό με τον οποίο προχωράει κάθε χώρα. Ευχαριστούμε για το πακέτο όσον αφορά την κατάσταση, πόσο προχωράει και που δείχνει την δέσμευση των χωρών αυτών υπέρ Τη ένταξή τους και την επιθυμία τους να τηρούν τα κριτήρια του Ελσίνκη. Το ο ρυθμός βέβαια εξαρτάται από την πρόοδο που κάνει κάθε χώρα. Και αυτό το αξιολογεί βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε όμως το Συμβούλιο να δώσει ένα σαφές μήνυμα όσον αφορά την πολιτική διεύρυνση. Ποιε είναι ακριβώ οι προϋποθέσεις της στήριξη των κριτηρίων από την κάθε υποψήφια χώρα ή την κάθε δυνάμει υποψήφια χώρα. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί των Δυτικών Βαλκανίων, για μας στη Βουλγαρία είναι ξεκάθαρο ότι ο μόνο σωστό τρόπος εξέλιξης των Δυτικών Βαλκανίων είναι τελικά να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό είναι ο δρόμο για την ανάπτυξη και την ευημερία και μην ξεχνάμε ότι οι χώρες αυτές ιστορικά, πολιτιστικά είναι μέλη της Ευρώπη. Δεν μπορεί λοιπόν να αποσιωπούμε από την άλλη μεριά και τα ανησυχητικά φαινόμενα που έχουμε στη Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχω πληροφορίες από τη Μακεδονία, λέει από την Σερβία, ανησυχητικές πληροφορίες για πολιτικές διώξεις που βασίζονται στην εθνική ταυτότητα. Και οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών πρέπει να λογοδοτήσουν για τις ε, κατηγορίες αυτές για τις υπόνοιες αυτές, γιατί εδώ φαίνεται ότι δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλες τις αρχές τις οποίες εμεί σεβόμαστε. Πάρε εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω κρατικά. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους Υπουργούς Εξωτερικών της Νοτιοδυτικής Ευρώπης, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων Φυσικά θέλω όλοι να προχωρήσετε και εγώ είμαι ε, αρμόδια για το θέμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ελπίζω ότι πολύ γρήγορα θα καταφέρει η Βοσνία Ερζεγοβίνη να σχηματίσει κυβέρνηση. Ε, πρόσφατα είχαμε συγκεκριμένα γεγονότα σε ό,τι φορά την θέση της Σερβίας απέναντι στη Ρωσία και τη, της ε, την περίπτωση του Σέσελ. Είχαμε διάφορες ε, εκδηλώσεις στα πλαίσια της επίσκεψης ε, Πούτιν στο Βελιγράδι, αλλά και κάποιες ασκήσεις ε, και γυμνάσια στα σύνορα Σερβίας-Κροατίας. Τα σύνορα Κροατίας πια δεν είναι μόνο εθνικά σύνορα, αλλά και κοινοτικά σύνορα. Ε, επίσης, οι δηλώσεις ως προς την διέξοδο της Σερβίας στη θάλασσα. Εμείς θέλουμε η Σερβία να βγει από την εντετερότητά της και να σταθεί στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού είναι πλήρες ε, υποψήφια χώρα και θέλει κάποια στιγμή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σίγουρα δεν θέλουμε εμεί να αποσταθεροποιηθεί η Σερβία με κανένα τρόπο. Θέλουμε απλώς να τηρηθούν και να γίνουν σεβαστές οι ευρωπαϊκές αξίες και αρχέ. Ε, ε, είπατε ότι θα πρέπει να επιστρέψει ο, ο Σέσελ στη Χάγη. Εμείς θέλουμε ρητά και κατηγορηματικά να κάνετε δηλώσεις υπέρ των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Και θέλουμε ε, να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τους ε, κοινοτικούς μηχανισμούς και να λάβετε υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα, λέει ο κύριος Πίτσουλα, να χαιρετήσω τους ε, Υπουργούς Εξωτερικών. Ε, δεν ε, υπάρχουν πολλές, ε, πολλοί ενθουσιασμό για τη διεύρυνση. Ε, α, δυστυχώς ήταν αρνητικές οι δηλώσεις του κυρίου Γιούνκερ. Βέβαια δεν πέθανε η διαδικασία της διεύρυνσης, αλλά κάπως επιβραβήθηκε φαίνεται ότι θα εφοδιάζεται με λιγότερα κονδύλια και χρηματοδότηση από ό,τι στο παρελθόν. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα Δυτικά Βαλκάνια για να συνεχιστούν οι προσπάθειες και οι μεταρρυθμίσεις. Ήταν πολύ καλή η πρωτοβουλία Λονδίνου και Βερολίνου να δοθούν ε, κίνητρα προς τη Βοσνία Ζεγοβίνη να συνεχίσει μεταρρυθμίσεις προς την ενταξιακή της πορεία. Βέβαια, όλε οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων χρήζουν υποστήριξη. Εγώ είμαι υπέρμαχος ε, τη ε, Ευρώπη, που φαίνεται, του τμήματο της Ευρώπης που ακόμη για καιρό δεν θα γίνει μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κροατία έχει σύνορα με τρει από τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι μόνο όταν μπουν και χώρε αυτέ των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος. Ε, έχουμε φυσικά σύνορα με μία χώρα που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτά που συνέβησαν στη Ιουγκοσλαβία. Αυτό που θέλω να πω στον Υπουργό Ντάτσιτς είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα για τον ΣΕΣΕΛ, για τον εγκληματία πολέμου, ουσιαστικά έκανε τη δική σας δουλειά, έκανε αυτό που έπρεπε να είχατε κάνει εσείς, δηλαδή να στυλτές και να καταδικάζει τις εμπριστικές και τις πολεμοχαρείς δηλώσεις του ΣΕΣΕΛ. Γιατί η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή ακριβώς βρέθηκαν ε, και υπό απειλή και υπονομεύθηκαν από τις δηλώσεις του ΣΕΣΕΛ και επειδή εσείς δεν κάνατε το δικό σας έργο να τις καταδικάσετε. Γνωρίζουμε ότι η απόλυση έγινε από τη Χάγη και ε, θα πρέπει να φροντίσει η Σερβία να κάνει δηλώσεις για το θέμα αυτό. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζω τη θέση που επικρατεί για τα Δυτικά Βαλκάνια. Προφανώς βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από κάποια χρόνια. Επίσης χαιρετίζω τους Υπουργούς Εξωτερικών που ήρθαν σήμερα εδώ ε, Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις τους. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, βεβαίως ε, διαφορετική είναι η πρόοδος που σημειώνουν τα κράτη αυτά στον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε υπέρ της διεύρυνσης όσον αφορά την πρόοδο της Βοσνίας Ερτσακοβίνης ε, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Ε, καλή πρωτοβουλία της ε, Γερμανία, να στηρίξει και χαιρετίζουμε την επίσκεψη του κυρίου Χάν και της κυρίας Μογκερίνη και εγώ θα επισκεφθώ αυτή την εβδομάδα την Βοσνία Ερσεγοβίνη. Ε, πρέπει να έχουμε μια νέα κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν για να αντιμετωπίσει τις ε, αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές αλλαγές για να αντιμετωπιστεί η οικονομική ανεπάρκεια και η διαφθορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω το εξής. Είναι αυτονόητο ότι στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τη διαδικασία διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ως Ρουμάνος πολίτης να βλέπω σήμερα χώρες που έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Και σκεφτείτε τι θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή προοπτική για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σήμερα κυρίως με μια ε, ασταθή, με ασταθείς εξελίξεις. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία στην περιοχή. Αυτή είναι προπόθεση για τη διεύνηση και επίσης και να υπάρχει και καλύτερος συντονισμός οποτεδήποτε γίνεται χρήση των ε, κοινοτικών κονδυλίων για τη δημιουργία υποδομών στην ενέργεια, στους σιδηρόδρομους, ε, στους αυτοκινητόδρομους. Το δεύτερο που θέλω να πω, ε, διμερείς συμφωνία στη διαδικασία διεύνηση, δηλαδή και από τα δύο κόμματα των χωρών, όπως σημαίνει στην Αλβανία και τη Μακεδονία, γιατί όταν υπάρχει μποϊκοτάρισμα αυτό είναι κίνδυνο και ζημιογόνο για μια χώρα. Επίσης να κρίνουμε τις χώρες από αυτά που επιτυγχάνουν και όχι από το παρελθόν τους. Κάποιες χώρες στην περιοχή θα πρέπει να παραιτηθούν από την προσπάθεια να αναφέρονται στην, ε, στο παρελθόν οποτεδήποτε ξεκινούν ε, τις ε, διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω τους Υπουργούς των Δυτικών Βαγανίων και θέλω να αναφερθώ στα όσα ρομαντικά ανέφερε ο Υπουργός της Φύρομ για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Όντως, ισχύει ότι η Ελλάδα προσπαθεί, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει και από τη γείτονα χώρα. Πρόσφατα είχα υποβάλει ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ονομασία τη Φύρομ και τη γλώσσα. Η απάντηση που πήρα από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι κακώς αναφέρεται η Φύρομ ως Μακεδονία και θα πρέπει να ισχύουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό είναι όντως σωστό, πράγμα το οποίο είδα ότι δεν συμβαίνει σήμερα στην Επιτροπή. Καταστρατηγείται δηλαδή από όλα τα μέλη η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και αναφέρεται η Φύρομ ως Μακεδονία. Γεγονός που είναι απαράδεκτο. Θέλω επίσης να τονίσω στον κύριο Υπουργό Εξωτερικών της Φύρομ ότι όσο η χώρα του καπηλεύεται την ιστορία και την ονομασία οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Ο ελληνικός λαός όμως δεν υπάρχει περίπτωση να συνηγορήσει για την είσοδο της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρος. Ε, προτείνω λοιπόν τώρα οι Υπουργοί των ε, Εξωτερικών να λάβουν το λόγο ε, με αντίστροφη φορά από ό,τι έγινε προηγουμένως. Αλλά επιτρέψτε μου πριν γίνει αυτό να κάνω την εξής παρατήρηση. Γνωρίζω από την ιστορία όλα αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Και παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι θαύμα το ότι στις 9 Μαΐου του 1950, πέντε χρόνια, μόλις πέντε χρόνια μετά τον δεύτερο, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρομπερ Σουμά έκανε σε εμάς τους Γερμανούς μία προσφορά ε, να συστήσουμε από κοινού την ΕΚΑΧ με βάση της, τη μη διακριτική μεταχείριση, με πλήρη ισότητα. Νομίζω λοιπόν ότι λαμβάνοντας υπόψη ε, τις ε, φρικαλαιότητες ε, του πρώτου και τελευταίου αποκριβισμού πολέμου αλλά και το ολοκαύτωμα, αυτό δεν το περίμενε κανείς. Αυτό ε, κατά τον 21ο αιώνα η επέτειος είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Το γεγονός ότι ο Ρόμπερ Σουμάν ποτέ δεν πήρε το Νομπέλ Ειρήνης για μένα εξακολουθεί να είναι και να παραμένει κάτι το πολύ οδυνηρό. Πέντε μόλις χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με όλα αυτά που έκαναν οι Γερμανοί. Και αν θέλετε αυτό είναι το κίνητρο της ευρωπαϊκής ανοποίησης. Το να πούμε ότι το παρελθόν δεν μας βοηθάει για το μέλλον. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι με μία μονοκοντιλιά ξεκάνουμε μία νέα αρχή. Και αυτό ισχύει και για τις διαδικασίες διεύρυνσης. Περί αυτού πρόκειται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να συμβάλλει στο να λύσει τα προβλήματα του παρελθόντος, αλλά το να τα καταστήσει περιτά βιώνοντας μία, μάλλον θέτοντας ένα κοινό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε όλοι. Και αυτή είναι μία διαδικασία που προφανώς και την εύχομαι και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτή είναι η βάση συμβίωσης γιατί αν θέλετε αυτή είναι η καρδιά της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης. Και αν το λάβουμε αυτό υπόψη μας τότε και οι επόμενες γενιές θα μπορέσουν να αποφύγουν όλα αυτά που κάναμε εμείς οι προηγούμενοι του παρελθόντος. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο πάνω σε αυτή τη βάση όλες οι πλευρές. Κανείς δεν αποκλείεται και αυτό δεν είναι προειδοποίηση προς μία πλευρά, όχι κάτι άλλο. Αφορά όλους, όλες τις πλευρές. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να σφυριλατηθεί η διαδικασία διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια που ήταν για αιώνες ολόκληρους θέατρο αιματοχυσιών και αιματηρών συγκρούσεων. Ελπίζω λοιπόν αυτή η διαδικασία, η διαδικασία των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων να μας οδηγήσουν στο σωστό δρόμο γιατί σας είπα αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία μπορούν να λειτουργήσουν όλα. Ich würde jetzt... Κατά τα άλλα, θα ήθελα να παρακαλέσω με αντίστροφη σειρά, όπως σας είπα, να δώσουμε το λόγο στους ε, Υπουργούς Εξωτερικών και αν έχω την καλοσύνη οι Υπουργοί Εξωτερικών να μιλήσουν για περίπου 4-5 λεπτά. Το θέμα δεν είναι ο καθένας εξ αυτών να μπει σε όλες τις λεπτομέρειες. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντάτιτς. Για μια και πριν ήμουν τελευταίος, τώρα θα είμαι πρώτος. Πραγματικά στην ομιλία μου δεν πιστεύω ότι ήμουν ούτε εχθρικός ούτε αλαζονικός, όπως με κατηγόρησε η κυρία Τόμασιτς. Νομίζω ότι η θέση σας ε, ε, σχετίζεται σε ένα πρόβλημα που έχει η, ε, η Σερβία. Έγινε πραγματικό τσίρκο γύρω από το Σέσελ, που ουσιαστικά το δικαστήριο της Χάγης το επέβαλε στη Σερβία. Δεν συμμετείχε η Σερβία στη διαδικασία αυτή φυσικά. Και ξέρετε, εμείς από πολιτική άποψη, η κυβέρνηση της Σερβίας, ο Πρωθυπουργός, εγώ και άλλοι υπουργοί δημοσίως ε, δήλωσαν ότι τέτοια πολιτική δεν έχει καμία πιθανότητα να τύχει υποστήριξη στη Σερβία αποκλείεται να υποστηριχθεί στη Σερβία. Κανένας φυσιολογικός άνθρωπος στη Σερβία δεν μπορεί σήμερα να στηρίξει μια τέτοια πολιτική σαν αυτή που παρουσιάζει ο Σέσελ. Δεν ξέρω, ίσως ε, αν ήσασταν στο Βελιγράδι ε, ε, και μάλιστα όταν συζητήσαμε στο Βελιγράδι με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομίζω ότι τα σαφίζει η θέση μας. Έγιναν δημόσιες δηλώσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κατάλαβε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να δίνουμε, να απολογούμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε. Έφυγε η κυρία Τόμασιτς, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, εγκατέλειψε την αίθουσα. Εγώ σέβομαι οποιονδήποτε ε, που ε, θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα της ε, Κροατίας. Αλλά όπως είπε κάποιος, κάθε χώρα έχει το σέσελ της. Και όπως ε, κάποιος είπε στην κροατική τηλεόραση, όποιος δεν αρέσει ε, η Κροατία ας σηκωθεί να φύγει. Τι είναι αυτό, αυτό είναι οι ευρωπαϊκές αξίες, αυτές είναι οι ευρωπαϊκές αρχές που θέλετε και εμείς να στενιστούμε. Δεν μπορώ να δεχτώ να λαμβάνω από την κυρία Τόμασιτς κήρυγμα και μαθήματα για τις ε, ευρωπαϊκές αξίες στη Σερβία. Δεν απελευθέρωσε η Σερβία το ΣΕΣΕΛ, δεν τον αποφυλάξει από τη Χάγη. Και μάλιστα σήμερα στη Σερβία ε, έγιναν ε, κοινά στρατιωτικά γυμνάσια της ε, Σερβίας, της Κροατίας, της Βουλγαρίας, της Ουρμανίας και της Μακεδονίας. Έχουμε στρατιωτική συνεργασία με όλες τις γειτονικές χώρες και είμαστε στρατιωτικά ουδέτεροι. Η Ρωσία δεν επηρεάζει τον πολιτικό προσανατολισμό της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πλένκοβιτς που είπε να κατηγορήσουμε τη ρητορική. Να είμαστε όμως σωστοί και δίκαιοι. Να καταδικάζουμε και να στυλιτεύουμε τέτοιες ρητορικές όπου και αν εκφωνούνται. Όχι μόνο να κοιτούμε τους γείτονες και τα του οίκου μας να κοιτάμε. Εμείς δεν, δεν μας αρέσει ούτε το κίνημα των ούστασης στην Κροατία, ούτε η εκστρατεία κατά του κυριλικού αλφαβήτου στην Κροατία. Και, εμείς, και εγώ όταν ήμουν Πρωθυπουργό. Δούλεψα πολύ και, κοπιά, και κόπιασα για την εξομάλυση σχέσεων με την Κροατία. Και κανένας δεν μας ενόχλησε τότε στην προσπάθεια γιατί δεν κοιτούσαμε προς το παρελθόν. είχαμε πολύ καλές συναντήσεις και στο Βελιγράδι και στο, στην Οπάτια και σε άλλες πόλεις και της Κροατίας και της Σερβίας. Και έχουμε πολιτική βούληση να προχωρήσουμε. Θέλουμε να πάμε προς τα μπρος. Δεν θέλουμε να παρεθοντολογήσουμε ούτε να παλινδρομήσουμε. Αυτά ως προς τις συζητήσεις Σερβίας και Κροατίας. Δεν είπα, κυρία μου, ότι η Σερβία διεκδικεί διέξοδο προς τη θάλασσα. Αστιεύτηκα και είπε ότι η Σερβία είναι η μόνη χώρα από την πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιουνίου που δεν έχει έξοδο στη θάλασσα. Το είπα αστειευόμενος. Γιατί αυτή η πρωτοβουλία αφορά την Αδριατική και το Ιόνιο και από η ιστορική άποψη είχε αυτή την ε, ιστορική επιθυμία η Σερβία. Αλλά γνωρίζουμε και δεν έχουμε καμία πρόθεση να βγούμε προς τη θάλασσα. Α, εσείς έχετε πρόθεση να έρθουν οι Σέρβοι προς τη θάλασσα, να βγει η Σερβία προς τη θάλασσα. Τι να σας πω. Θα σας πω το εξής. Εγώ Ε, η Κροατία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνει υπόδειγμα, παράδειγμα προ μίμηση για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Δεν χρειάζεται να αγαπιόμαστε, αλλά τουλάχιστον να κοιτάμε προ το μέλλον. Να ζητούμε την πρόοδο και όχι να καυγαδίζουμε. Εύκολο είναι ο καυγάς, εύκολο είναι να μαλώνουμε. Εμείς καταδικάζουμε κάθε πολιτική που υπονομεύει ή ε, απειλεί την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Εθνικιστικές δηλώσεις, νεοναζιστικές ε, ε, που ακούστηκαν και στη Σερβία με τους ΕΣΕΛ και στην ε, Κροατία. θυμάστε τι έγινε στο γήπεδο με, τις, με τη σημαία και τη Μεγάλη Αλβανία. Υπάρχουν τέτοιες εθνικιστικές εξάρσεις παντού στην περιοχή. Παρακαλώ όμω, κοιτάξτε και αναγνωρίστε τη τεράστια πρόοδο που πραγματοποιήσαμε τον τελευταίο καιρό. Δεν ήταν εύκολο και εγώ είμαι έτοιμο να προσπαθήσω ακόμη περαιτέρω για την ομαλοποίηση των σχέσεων και με την Κροατία. Και θα πρέπει με όλους ε, να φροντίζουμε, όποιος και αν είναι στην εξουσία, να βελτιώνουμε τις σχέσεις μας. Δεν διαλέγει ο καθένας που γεννιέται, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Μπορούμε όμως να δουλέψουμε για το παρόν και το μέλλον. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των Βαλκανίων σε τελική ανάλυση, ότι υπάρχει αυτή η πολυμορφία και η πολυεθνότητα, αλλά δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλον. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο κύριος Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ανταλλάσσουμε απόψεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Και ευχαριστώ πολύ για τα θετικά σας λόγια. Δύο πράγματα θέλω να σχολιάσω σύντομα. Πρώτον, ε, ρωτήσατε για τις μεταρρυθμίσεις μας. Αφού προχωρήσαμε σε συνταγματικές ε, τροποποίησεις, συζητήθηκε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων στο Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα περάσει κιόλα. Ήδη έχει μπει στο αυλάκι. Πρόκειται για το δικαστικό τομέα, την ανεξαρτησία του, για το γραφείο εισαγγελέα, για το στοματικό δικαστήριο, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαστών και ένα πακέτο κατά της διαφθοράς για το χρηματισμό, για τα λόμπις, τις ε, ομάδες συμφερόντων δηλαδή και το κώδικα διοντολογίας των βουλευτών. Είναι ένα πακέτο λοιπόν πολύ ουσιαστικό. Και βγαίνει βέβαια από τη δράση μας όσον αφορά τα κεφάλαια 23 και 24. Αυτό το πακέτο νόμων θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για μας για να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και να δείξουμε πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στις μεταρρυθμίσεις μας. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη ερώτηση, είχε να κάνει με τους Ρώμα και την ένταξή τους στην κοινωνία. Μία από τις προτεραιότητάς μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αυτό και έχουμε πάρει διάφορα μέτρα για να το πετύχουμε. Πρόκειται για την εκπαίδευση, για την αγορά εργασίας, που έχουμε πετύχει αξιοπρεπείς επιτυχίες. Υπάρχει και ο μηχανισμός αξιολόγησης βέβαια της Επιτροπής και του Συμβουλίου και υπάρχουν και κοινοβουλευτικές επιτροπές που κάνουν το ίδιο. Μαζί λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών θα συνεχίσουμε να προχωρούμε και να κάνουμε βήματα και σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα αγγλικά μίλησα την πρώτη φορά, τώρα θα μιλήσω γερμανικά, γιατί και ο κύριος Παπόσκη και, και εγώ ερχόμαστε μετά από μια συνάντηση που είχαμε για την φραγκοφωνία, τη γαλλοφωνία. Το κοσυφοπέδιο αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητη χώρα. Την επόμενη φορά θα μιλήσω γαλλικά. Τώρα όμως θα μιλήσω γερμανικά. Κυρίες και κύριοι, για μένα πρέπει να ξέρετε ότι είναι μεγάλη χαρά που μπορώ να έρθω εδώ και να απαντήσω σε ερωτήσεις που τέθηκαν όσον αφορά το κοσυφοπέδιο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να το δω στα ερωτήματα που ετέθησαν. Πιστεύω ότι το θεμελιώδης ερώτημα είναι το, ε, τι μορφή θα έχει λάβει η περιοχή μετά από πέντε χρόνια. Δηλαδή τι μορφή θα έχουν λάβει τα Δυτικά Βαλκάνια. Παλαιότερα το σκέχω σκεφτεί αυτό το πώς μπορούσε, θα μπορούσε να διαμορφωθεί ε, το καθεστώς ε, στην περιοχή. Εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στρέφει προς εμάς την ε, προσοχή μας. Όμως, αν κατά τα επόμενα πέντε έτη η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται πραγματικά για τη σταθερότητα, Νομίζω ότι η περιφερειακή σταθερότητα πρέπει να επικρατήσει και στα Βαλκάνια και πρώτα απ' όλα πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει σταθερότητα. Νομίζω λοιπόν ότι όσον αφορά στα Βαλκάνια η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κατά την άποψή μου δεν πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση της ε, διεύρυνσης αλλά της ε, σταθεροποίησης. Δηλαδή δεν νομίζω ότι στόχος είναι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία ή η Τουρκία να υπάρχουν πιο πολλές στενές σχέσεις με τις χώρες που παραδοσιακά ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, Θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο σημαντικές ε, περιφερειακές ε, προκλήσεις και οι εξελίξεις στα Βαλκάνια θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις προκλήσεις αυτές. Η πρώτη πρόκληση έχει να κάνει με τα ανοιχτά διμερή θέματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσφοπεδίου. Εμείς από δικής μας πλευράς είμαστε πρόθυμοι ε, σε ένα χρονοδιάγραμμα τριών έως πέντε ετών να ρυθμίσουμε όλα τα ανοιχτά θέματα με τη Σερβία και να υπογράψουμε συμφωνία ειρήνης η οποία θα οδηγήσει και σε συμφωλίωση των δύο λαών. Ανεξάρτητα όμως από την διαδικασία ομαλοποίησης ανάμεσα στο κοσφοπέδιο και τη Σερβία υπάρχουν και άλλα ανοιχτά θέματα στην περιοχή που δεν θέλω να τα δείξω σκόπιμα γιατί έχω εδώ τους συναντέλφους μου που παρίστανται. Το δεύτερο θέμα που έχει σχέση με τις περιφερειακές αυτό έχει σχέση με την διακρατική συμφιλίωση, με την έλλειψη οικονομικών σχέσεων. Έχει σχέση το δεύτερο αυτό και με την έλλειψη επενδύσεων, κυρίως όμως έλλειψη κράτους δικαίου ελλειπής προστασία των μειονοτήτων, ε, της ελευθερίας του τύπου, κάτι το οποίο νομίζω ότι έδειξαν ε, αρκετοί συνάδελφοι. Όσον αφορά τώρα στο κοσφοπέδιο, θέλω να σας πω ότι ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα κατά τα επόμενα έτη να συνεχίσουμε τη διαδικασία σταθεροποίησης του νεόκοπου κράτους μας. Εν τω μεταξύ, μας έχουν αναγνωρίσει 108 κράτη. Είμαστε μέλος σε διάφορους ε, περιφερειακούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς. Το Κωσυφοπαίδιο είναι κράτος και θα παραμείνει κράτος. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν έχουν ε, αναγνωρίσει ακόμα το κοσυφοπαίδιο να τοποθετηθούν επ' αυτού και να το αναγνωρίσουν. Αυτό θα ενδυναμώσει και την Ευρώπη και το κοσυφοπαίδιο. Και παράλληλα, ως πολιτικός του κοσμοπεδίου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω κατά τα επόμενα έτη να δώσετε τη δυνατότητα κατάργησης θεωρήσεων στους πολίτες μας. Εφέτος, ελήφθη μία απόφαση για τη Μολδαβία. Πλέον καταργήθηκαν οι θεωρήσεις από και προς τη Μολδαβία. Και θεωρώ ότι την προηγούμενη Κυριακή, αν δεν είχε γίνει αυτό, θα ήταν τελείως διαφορετικό το εκλογικό αποτέλεσμα ε, στη Μολδαβία. Το ίδιο ισχύει και για το Κοσμοπέδιο. Χρειαζόμαστε την ισχυρή πολιτική βούληση έτσι ώστε οι πολίτες μας ε, κατά τα επόμενα έτσι και του χρόνου να μπορούν να ταξιδέψουν ε, ελεύθερα στα κράτη Σέγγεν. Κύριε Μπροκ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που με προσκαλέσατε με τους συναντέλφους μου από την περιοχή σε αυτή την συνάντηση και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα εθνικά κοινοβούλια για την αμέριστη υποστήριξη που προσφέρουν στο Κοσφοπέδιο. Ο πρόεδρος δυστυχώς ομιλεί εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουν υποθεί τα πιο σημαντικά πράγματα και το πιο σημαντικό που είπαμε είναι ότι δεν διορθώνουμε τις ιστορικές αδικίες, αλλά προσανατολιζόμαστε στο μέλλον. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, το πιο σημαντικό εδώ θα ήταν ότι όταν μας ενδιαφέρουν οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές μάλλον και οι ευρωπαϊκές αξίες, θα πρέπει τη μεγαλύτερη ενέργεια να μην τη δώσουμε στο να βγάλουμε τη μακεδονική γλώσσα ή την ε, μακεδονική εθνικότητα από τα κείμενα, αλλά να επικεντρωθούμε στα δημοκρατικά δικαιώματα, σε πράγματα που ενδιαφέρουν πιο πολύ τον κόσμο. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να στηρίξουμε τις διαπραγματεύσεις που αποτελούν το μέσο ώστε χώρες μέλη να έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στις μεταρρυθμίσεις. Και μεταρρυθμίσεις χρειάζονται. Είναι γεγονός αυτό για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Και αυτό δεν γίνεται στα πλαίσια του να βεβαιωθούμε για τις μεταρρυθμίσεις δυστυχώς, αλλά για να το χρησιμοποιήσουμε για άλλους λόγους. Μιλάω βέβαια για την Μακεδονία λέει Όχι γιατί, το λέω αυτό όχι γιατί έχει κρατήσει υπερβολικά πολύ η διαδικασία, γιατί έχουμε εμεί στηρίσει όλες τις προδιαγραφέ, αλλά υπάρχει συμφωνία γι' αυτό. Και υπήρξαν ε, πολιτικοί που λένε και εξακολουθούν και σήμερα να λένε ότι αν δεν υπάρξει αποδεικτή διαδικασία για να ενταχθεί στην Ευρώπη η Μακεδονία θα δημιουργηθούν ταραχές οι οποίες ή προβλήματα τα οποία δεν θα μπορέσουν να λυθούν εύκολα. Αυτό είναι κάτι όμως που ανήκει στο παρελθόν και δεν πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε περισσότερο εκεί. Χρειαζόμαστε όμως συνένεση. Ίσως για να διδαχτούμε για το συσχετισμό δυνάμεων και για το ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να βάλουν προϋποθέσεις στο τραπέζι, όρους, πείτε τους όπως θέλετε, που να μην ευθαγραμματίζονται πάντα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην τηρείται πάντα το κράτος δικαίου. Και χαίρομαι που το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το Διεθνές Δίκαιο αναφέρθηκαν. Γιατί είναι σαφέστατα. Πρόκειται για Διεθνές Δικαστήριο που λέει ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει ένα άλλο όνομα από αυτό το οποίο δημοκρατικά έχει επιλέξει μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα. Και από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έρχεται καμία άλλο, άλλη υποχρέωση πέρα από αυτές τις οποίες αναφέρει το ψήφισμα. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις καλές σχέσεις που έχουμε με την Ελλάδα, τη γείτονά μας νοτίως, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε κοινέ πολιτικές κοινούς μάλλον πολιτικούς και στρατηγικούς στόχους. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για την εσωτερική κατάσταση. Και για να μην χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα, θέλω να είμαι σαφής. Έχουμε διαφορές για πάρα πολλά πράγματα, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Αλλά έχουμε στην Μακεδονία συμφωνία με πολιτικές, θρησκευτικέ ε, και άλλες κοινότητες όσον αφορά το μέλλον μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό ακριβώς δεν θέλουμε να χρησιμοποιείτε το επιχείρημα που λέει ότι εφόσον δεν λύνεται το, όνομα, το θέμα του ονόματος η Μακεδονία πρέπει να μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκαν διάφορες πραγματικότητες εδώ και πράγματι και εμείς στα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να συνειδητοποιούμε την πραγματικότητα. Η πρώτη πραγματικότητα είναι ότι κανείς δεν θα χαρεί άμα ακούσουμε ότι σήμερα οι εξωχώρες των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μια άλλη πραγματικότητα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι αν δεν έχουμε ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό μέλλον, μπορεί να χάσουμε ιστορικές ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας. Κάθε μία από τις αλλαγές που έχουν γίνει στο παρελθόν, τις τελευταίες δεκαετίες δηλαδή, μετά την ε, λήξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Δεύτερο, τη σχέση μας με τον κομμουνισμό κτλ. που βγήκαμε από τον κομμουνισμό, όλα αυτά έγιναν με αίμα και δάκρυα. Είναι η πρώτη φορά που η μετατροπή της κοινωνίας μας ευρωπαϊκή μπορεί να γίνει χωρίς τέτοιες θυσίες. Μην το ξεχνάμε αυτό, μην βγάζουμε τα πράγματα από το ιστορικό τους πλαίσιο. Πρέπει για να αποδείξουμε και εμείς ότι ο κύριος Σούμερ και ο κύριος Μονέ είχαν δίκιο με αυτά που είπαν, ότι πρέπει να τηρούμε τις αξίες, αξίες που λένε ότι όλοι έχουμε αξιοπρέπεια και δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και ο συνάδελφος Χότζεφ, αποφάσισα να αλλάξω γλώσσα στη δεύτερη μου παρέμβαση. Μπορεί κάποιοι να κέρδισαν από τη διάλυση της Ιουκοσλαβίας, αλλά νομίζω τελικά πολύ βγήκαμε χαμένοι. Όλοι χάσαμε πάρα πολλά. Αλλά ένα από τα θετικά είναι ότι μέσα σε μία νύχτα γίναμε πολύγλωση. Ξαφνικά, ενώ δεν ε, μάθαμε στο σχολείο, ξαφνικά μάθαμε να, ε, βρεθήκαμε να μιλάμε πέντε γλώσσες. Μαυροβουνικά, βοσνιακά, σερβικά, κροατικά. Εγώ μιλώ λοιπόν κροατικά που είναι μια από τις πολύγλωσσοι. γλώσσες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να ακούσω τη γλώσσα μου, τα βοσνιακά, ε, ελπίζοντας ότι κάποια μέρα θα γίνουν και τα βοσνιακά επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηρέμησε Ήβιτσα. και εσείς από την περιοχή είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ας α, ε, ε, είμαστε είτε όπως είμαστε μια χώρα, τώρα είμαστε πολλές χώρες χωρίς πόλεμο όμως, ανέμακτα, γιατί όλοι περιμένουμε στην αίθουσα αναμονής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν θα μιλήσω για το Σέσελ. Όταν μπήκα κάποιος με ρώτησε τι είναι αυτό εδώ στο πέτο σου, ε, ε, είπα μια και το, το θέμα είναι ο Σέσελ, εγώ θα φορέσω κάτι που ακριβώς δείχνει πόσο ε, βάναυσο παράδειγμα ήταν η πολιτική του Σέσελ και έβαλα το σήμα της Ρεμπρένιτσα. Και ε, σίγουρα ε, εδώ είναι το σύμβολο μιας ιδεολογίας και το σύμβολο των παθών που προκάλεσε αυτή η ιδεολογία. Και μακάρι να βρεθούμε όλοι στην ε, Σρεμπρενίτσα για να διδαχθούμε κάτι από αυτά, από την ιστορία και από το που οδήγησε μια ιδεολογία σαν αυτή του Σέσελ. Πάντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δώσετε να συναντηθούμε εδώ και να απαντήσω και σε ορισμένε ερωτήσεις. Η κατάσταση στη Βοσνία Ριζαγοβίνη πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αργά αλλά σταθερά. Καλύτερα όμως αργά προς τη σωστή κατεύθυνση, το καλό αργία γίνει, παρά γρήγορα προς τη λάθος κατεύθυνση. Πάμε προς τη σωστή πορεία, προς τη σωστή άγουσα και ελπίζω, ίσως όχι μέχρι τα τέλη του έτους, αλλά στην αρχή του επόμενου έτους να σχηματιστεί η κυβέρνηση και η πρωτοβουλία που ξεκίνησε, όπως θέλετε πείτε την, του Λονδίνου και των Βερολίνου, των Βρυξελών. Το θέμα είναι να μείνει κάποιο στίγμα από αυτή την πρωτοβουλία και να είναι πρωτοβουλία για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρθηκε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να γίνει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, πανευρωπαϊκή, όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να... Και φυσικά καλό θα ήταν να τύχει της υποστήριξης και της άλλης όχθης του Ατλαντικού. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία ως πλατφόρμα για περαιτέρω πρόοδο, για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και μετά να δημιουργήσουμε την κυβέρνηση. Και όχι να σχηματίσουμε πρώτα την κυβέρνηση χωρίς να έχουμε προηγουμένως την πλατφόρμα για τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό και είναι πολύ ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη η πρωτοβουλία και πιστεύω ότι μας δίνει πραγματικά μια σοβαρή ευκαιρία για πρόοδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, επιρροή της Ρωσίας ή του ριζοσπαστικού Ισλάμ ε, στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κάποιος είπε ότι όταν δημιουργείται ένα κενό στην περιοχή, το κενό αυτό δίνει την εντύπωση ότι η πορεία προς τον ΝΑΤΟ και η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χρονοβόρα και πολύ μακριά. Οπότε αν δημιουργηθεί αυτό το κενό ως προς τις βλέψεις του για τον ΝΑΤΟ και την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιο θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το κενό. Ελπίζω όχι η Ρωσία και ελπίζω όχι οι τζιχαντιστέ. Ελπίζω να μην δημιουργηθεί το κενό και να μην τεθεί ένα αμφιβόλο η ευρωπαϊκή μας πορεία, η πορεία προ τον ΝΑΤΟ. Οποιοδήποτε, ε, η, η Τουρκία, η, το Ιράν, η Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω κανένας να μην έχει πρόβλημα με την ενταξιακή μας προπτική. Το θέμα είναι να μην έχει κανένα στη Βοσνία πρόβλημα με την ενταξιακή μας προπτική. Θέλω να υπάρχει απόλυτη συμφωνία και συνένεση στη Βοσνία για την ευρωπαϊκή μας πορεία όλες οι εθνότητες, οι στατικές, όλες οι μειονότητες ε, να είναι υπέρ της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης ομοφωνία για το ΝΑΤΟ. Δεν νομίζω κανένας να αμφισβητεί σήμερα την πορεία μας είτε προς τον ΝΑΤΟ είτε στην, προς τον Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει απόλυτη σύμπνοια ως προς αυτό. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσω στα αγγλικά, γιατί το σύνταγμά μας είναι το σύνταγμα του Dayton που το έχουμε στα αγγλικά, που δεν το έχουμε ακόμη μεταφράσει, γιατί δεν έχουμε συμφωνήσει πώς θα πρέπει να μεταφραστεί στα βοσνιακά ή σερβικά ή κροατικά ίσως θα πρέπει να έχουμε ένα νέο, να κάνουμε μια αναθεώρηση του συντάγματος και να έχουμε μια νέα συνταγματική ένωμη τάξη. Γιατί είχαμε κάποιες αρνητικές ε, αξιολογήσεις, τώρα θέλουμε μια θετική αξιολόγηση. Τώρα, ως προς την ερώτηση της Μαρή Λουίς για τον Ντόντικ και το δημοψήφισμα. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να γίνει δημοψήφισμα. Δεν νομίζω ότι κανένας είναι τόσο παλαβός για να ζητήσει κάτι τέτοιο. Μόνο ένας Θεότρελος θα μπορούσε να ζητήσει κάτι τέτοιο δημοψήφισμα για απόσχεση που είναι κατάφορη παραβίαση του συμφωνία της συμφωνίας του Ντέιτον. Άλλωστε, οποιαδήποτε παραβίαση της, της συμφωνίας Dayton θα προκαλέσει άμεση επέμβαση της διεθνούς κοινότητας, γιατί κανένας δεν έχει συμφέρον να παραβιάσει και ελπίζω και έχει και φιλοδοξία να παραβιάσει τη συμφωνία του Dayton, παρόλο που μπορεί να γίνονται κάποιες δηλώσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να κάνει τη δουλειά του και το καθήκον του. Και πάνω απ' όλα να κάνει αυτό που είναι σημαντικό για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γιατί άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο ειρηνική συνύπαρξη και αμοιβαίου σεβασμού. Δεν θα πρέπει ο καθένα να χρησιμοποιεί αρνητικού χαρακτηρισμού για το γειτονά του ή να τον βλέπει με αρνητικό φω. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τι διαφορέ μα. Και αν δεν το καταφέρουμε αυτό στη Βοσνία Ερζεγοβίνη πώς ε, ε, θα μας δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δεχτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη στις διαφορές, στα διαφορετικά. Βλέπετε, Άξε επέτρεψε στον εαυτό μου να μακρηγορήσω για να δω πώς ακούγονται τα βοσνιακά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τελευταία πρόταση μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους υπουργού Εξωτερικών για το ότι ανέχτηκαν τη συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών και συζήτησαν μαζί μας. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι για μας, για τους περισσότερους από εμάς, είναι σαφής η τοποθέτησή μας ως προς τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, είναι σαφές ότι θα πρέπει κάπως ε, να ξεπεραστούν οι διμερείς διαφορές ε, στα διάφορα κράτη. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω όλα αυτά και ευελπιστώ αυτή η διαδικασία να έχει αίσιο τέλος και σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Όσον αφορά τώρα το θέμα του, του ποινικού δικαστηρίου, εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν έχω καταλάβει τελικά τι κάνει αυτό το ποινικό δικαστήριο, αν κάνει κάτι. Φαντάζομαι αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολλούς. Πάντως είναι ένα θέμα ε, που θα μας απασχολήσει ανεξάρτητα από αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση του Σέσελ. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους αντέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζητήση αυτών των τελευταίων δύο ημερών. Εγώ προσωπικά τις συζητήσεις αυτές τις βρήκα ιδιαίτερα επικοδομητικές και ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς από αυτού. Θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε μια τέτοια συνάντηση και να ξανασυναντηθούμε μια επόμενη φορά έχοντας υπόψη την συνάντηση του Ιουνίου, συνάντηση άμυνας, να καλέσουμε το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ίσως κατά το Φεβρουάριο, κάπου εκεί. Δεν ξέρω αν ε, θα τα καταφέρετε να έρθετε, αλλά μπορείτε να σημειώσετε αυτή τη συνάντηση του Φεβρουαρίου. Σήμερα το απόγευμα συνεχίζεται η συνεδρίασή μας και όποιος θέλει ευχαρίστως μπορεί να συμμετάσχει. Αν θέλετε να σας ε, αναφέρω και τα σημεία της σημερινής διάταξης. Στις 3 η ώρα θα έχουμε τη συζήτηση με τον κύριο Μικάλ Κοντοκόρφσκι και κατόπιν στις 4 ε, με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου και στις 5 η ώρα ανταλλαγή απόψεων με τον Μπερναντίνο Λεόν σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη. Αν κάποιο από εσά ενδιαφέρεται για κάποιο από αυτά τα θέματα, πολύ ευχαρίστω να έρθει να παρακολουθεί τις συνεδρίες. Αν όχι, καλή επιστροφή στις πατρίδες σας, καλό μεσημέρι. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα και αν δεν δω σύντομα κάποιους από εσάς, σας εύχομαι και καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που ήρθατε.